Nein, nein, nein. Dear colleagues, dear guests, uh, dear uh, visitors uh, at... Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 9 και 5. Πρέπει να αρχίσει η Επιτροπή μας, η συνεδρίασή μας. Χαιρετίζω τους συναδέλφους που είναι ήδη παρόντες. Πρώτο θέμα, Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν προτάσεις τροποποίησης. Όχι, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Με μία τροποποίηση. Το τελευταίο σημείο 24 πρέπει να αναβληθεί γιατί ο εισηγητής μας δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Ωραία, συμφωνείτε και με αυτό βλέπω. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών. Ω συνήθω, αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση, θα θεωρηθεί ότι είναι χρήθησαν. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Ο 15ος γύρος των συνομιλιών στη Γενέβη και κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουν να καταλήξουν φέτος οι εργασίες. Αυτό νομίζω ότι είναι καλό ε, μήνυμα και για το πολυμερές σύστημα. Ορισμένοι θεωρούσαν ότι στην ουσία έχει εκπνεύσει, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι, ακόμη ζει και λειτουργεί. Επίσης θα συζητήσουμε για την προστασία των επενδύσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Μιανμάρ. Και ο Επίτροπος και οι Υπουργοί θα συζητήσουν την προστασία των επενδύσεων. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Σημείο 4. Συνεχιζόμενοι τριμερείς διάλογοι. Κατέληξαν δύο τριμερείς διάλογοι και ευτυχώς λοιπόν έχουν καταλήξει οι δύο που είχαμε και δεν υπάρχουν συνεχιζόμενοι τριμερείς διάλογοι. Και αυτό είναι ευχάριστο και για την γραμματεία γιατί είναι πολλή δουλειά η τριμερής διάλογοι. 5, το σημείο 5, πολύ ενδιαφέρον νομοθέτημα και σημαντικό Ιδιαίτερα γιατί είμαι ο εισηγητής. Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου. Εγκρίναμε τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση το Μάρτιο του 2014 και ξεκίνησε έκτοτε ο τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και συμφωνήσαμε σε ένα κείμενο αλλά το Συμβούλιο δεν απεδέχθη το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου, παρά το ότι η Προεδρία ήταν υπέρ. Ιδιαίτερα συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο και αντιμετώπιση των κατεξοδότηση ε, και εκτελεστικών πράξεων δημιούργησαν προβλήματα. Δεν είχαμε όμως επίσημη αντίδραση του Συμβουλίου. Οπότε το θέμα παρέμενε εκρεμές. Και μετά την διοργανική συμφωνία, την κατάληξη τον περασμένο Δεκέμβριο σε διοργανική συμφωνία, μπορέσαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη διοργανική συμφωνία και για το θέμα αυτό Η Επιτροπή μας ενέκρινε το κείμενο την 21η Απριλίου και το Συμβούλιο κατόπιν μετά από δύο μήνες στις 16 Ιουνίου ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δική μας ανάγνωση, δηλαδή πολλές φορές μας παίρνει πολύ χρόνο μέχρι να υπάρξει πρόοδος. Προτείνω λοιπόν τώρα η ΙΝΤΑ να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες γιατί είναι αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου και πολλά από τα σημεία των απόψεων του Κοινοβουλίου έχουν συμπεριληφθεί και τα διοργανικά θέματα ρυθμίστηκαν από τη διοργανική συμφωνία. Προτείνω λοιπόν να εγκριθεί χωρίς τροπολογίες. Θέλει κανείς το λόγο επ' αυτού? Όχι. Α, τι έκπληξη. Ούτε η Επιτροπή θέλει το λόγο. Απίστευτο. τόσο σημαντικό θέμα κοσμοϊστορικής σημασίας και κανείς δεν θέλει το λόγο. Εν πάση περιπτώσει. Προθεσμία για τροπολογίες σήμερα 6 ώρα το απόγευμα. Γιατί θέλουμε να ψηφίσουμε επ' αυτού για αυτό το θαυμάσιο θέμα λοιπόν αύριο. Ωραία. Οπότε περνάμε στο 6. Γνωμοδότηση για την Ήτρε. Για τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για διακυβερνητικές συμφωνίες και μη δεσμευτικά μέσα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και η κατάργηση μίας απόφασης. Και δίνω απευθείας το λόγο στον κύριο Μπέρντζεν, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Είναι γνωμοδότηση για μια εργασία που γίνεται στην Ήτρε όπου είμαι και μέλος. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη είναι υπέρ της διατήρησης του status quo, αλλά όπως και οι συνάδελφοί μου στην Ήτρε προτείνω η Επιτροπή μας να στηρίξει την Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνίες με τρίτες χώρες για θέματα ενέργειας που δεν συμμορφούνται με τον ενωσιακό νόμο. Υπάρχει απόφαση που λέει ότι αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να αξιολογούνται μετά την υπογραφή τους, αλλά η Κομισιόν προτείνει να αλλάξει αυτό, ούτως ώστε να αξιολογούνται πριν την ε, κατάληξη σε τελικό κείμενο, γιατί είναι δύσκολο κατόπιν, όπως έχουμε δει ε, από την πείρα μας, να υπάρξει αναδιαπραγμάτευση μετά την υπογραφή τους. Αυτό έχει έννοια, είναι σημαντικό ε, τα κράτη-μέλη να δρουν από κοινού έναντι τρίτων χωρών. Βλέπουμε αυτή τη δυναμική με την εμπορική λογική. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι από κοινού 28-27 από ότι μεμονωμένα. Πρέπει να στηρίξουμε την Κομισιόν, να έχουμε εξάντε αξιολόγηση των διακυβερνητικών συμφωνιών. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να στηρίξουμε το πεδίο εφαρμογής που προτείνει η Κομισιόν να καλύπτει και μη δεσμευτικές συμφωνίες και μη δεσμευτικά μέσα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έχω κάποιες προτάσεις αλλαγή στο κείμενο. Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Θα έλεγα να καταστήσουμε πιο ισχυρή τη σύνδεση με την Ενεργειακή Ένωση και τις ενωσιακές αρμοδιότητες όπως κοινή εμπορική πολιτική και να συμπεριλάβουμε και συμφωνίες στις ε, ε, οποίες ε, καταλήγουν διάφορες επιχειρήσεις εάν παίζουν ρόλο οι κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να κρύβουμε διακυβερνητικές συμφωνίες με έξυπνες ε, δομές για την ε, ιδιοκτησία. Υπάρχει μία επιχείρηση που κατά 58,1% είναι ιδιοκτησία του ε, δανέζικου κράτους. Θα έπρεπε λοιπόν να θεωρηθεί μια συμφωνία αυτής της εταιρεία ως διακυβερνητική, διότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες μας, για να επιτύχουμε το στόχο της Ενεργειακής Ένωσης που είναι η ασφάλεια προμηθειών. Γιατί ορισμένες τέτοιες συμφωνίες ε, περιέχουν άρθρα τα οποία αντιβαίνουν τους στόχους μας ε, και την νομοθεσία μας. Η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αποφύγουν τις παγίδες, να τα καθοδηγήσει καλύτερα. Είναι προς το συμφέρον των συμπολιτών μας, αλλά και των επενδυτών γιατί θα έχουν περισσότερη επενδυτική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος, κύριε Μπένσεν. Και τώρα η σκιώδη. Ντάντι, σοσιαλιστής. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συγγνώμη που ήρθα με καθυστέρηση, αλλά είχα πολύ δουλειά το πρωί. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησής του οι τροπολογίες του είναι αποδεκτές εν μέρη για την τροποποίηση αυτής της απόφασης για έλεγχο εκ των προτέρων εκ μέρους της Επιτροπής συμφωνώ με αυτή την διτή προσέγγιση που προτείνει. Αφενός δηλαδή να διευκολύνουμε μια μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών στο τομέα της ενέργειας ενισχύοντας τον ρόλο της Κομισιόν ως θεματοφύλακα των διακυβερνητικών συμφωνιών τη Ένωση, χωρίς να επιστρέφουμε στην ουσία και αφετέρου να διασφαλίσουμε την απαραίτητη εχεμήθεια στις διαπραγματεύσεις τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα τομέα όπου η αρμοδιότητα εμπίπτει κυρίως στις χώρες μέλη και έχουμε να κάνουμε με συμφωνίες. Η Κομισιόν θα πρέπει να διασφαλίσει την διαχείριση των ε, πληροφοριών που αναφέρονται σε ευαίσθητες από τις χώρες μέλη, όπως εξάλλου σημαίνει σήμερα με τα έγγραφα διαπραγματεύσεων της Κομισιόν στι εμπορικέ συμφωνίες. Θα είναι σημαντικό η αξιολόγηση που θα δώσει η Κομισιόν να περιοριστεί στη διασφάλιση της συμφωνίας με το δίκαιο της Ένωσης και αυτό θα πρέπει να γίνει έγκαιρα και πρόθεσμα για να μην δημιουργηθούν φραγμοί και εμπόδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την σύναψη της συμφωνίας. Θεωρώ επίσης ότι η δυνατότητα η Κομισιόν να παράσχει βοήθεια σε χώρες μέλη πρέπει να εξαρτάται από την της κάθε χώρας μέλου. Καταλήγοντας, στηρίζω την πρόταση της ε, Κομισιόν και συμφωνώ ότι κάποια μέρη της πρότασης που αφορούν τους χρόνους ή τον εμπιστευτικό χαρακτήρα πρέπει να ισχυθούν και γι' αυτό θα καταθέσω τροπολογίες. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα προς μια ένα μεγαλύτερο συντονισμό και εναρμόνιση στον τομέα της ενέργειας. Εν βέβαια μιας μεγαλύτερης ε, συνοχής, ενεργειακής πολιτικής, πολιτικής, εσωτερικής αγοράς ενέργειας και ανταγωνισμός σε αυτό το βασικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς. Ο κύριος Ζάραντιλ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά όχι μόνο την ε, ενεργειακή πολιτική της Ένωσης, αλλά και άλλες ε, πολιτικές ε, της νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα η εσωτερική αγορά, οι δημόσιες προμήθειες και το εμπόριο. Συνεπώς η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας είναι πολύ σημαντική. Δεδομένων κάποιων ε, διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή ε, ένα ενεργειακό κεφάλαιο στο πλαίσιο της συμφωνίας ε, TTIP με τις Φιλιππίνες. Πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχει και μια πολιτική ευαισθησία Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών σε ποιο βαθμό θα αυξηθεί η διαφάνεια και σε ποιο βαθμό θα συμμετέχει άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, διαφορετικές αυτές απόψεις και να μπορέσουμε να βρούμε έναν βιώσιμο ε, συμβιβασμό μεταξύ των κρατών μελών. Για το σχέδιο γνωμοδότησης, θα ήθελα απλώς δύο σημεία να επισημάνω. Αν κατάλαβα καλά, η άποψη του εισηγητή είναι ότι η προτινόμενη απόφαση δεν θα έπρεπε να δημιουργεί υποχρεώσεις σε σχέση με τις συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικών φορέων, όμως θα εξακολουθήσει να ισχύει για διακυβερνητικές συμφωνίες, ε, δηλαδή συμβάσεις ε, και συμφωνίες μεταξύ εταιριών θα καλύπτονται από διαφορετικά ε, διαφορετική απόφαση. Αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ. Συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να κοινοποιούν τέτοιου είδους ε, συμφωνίες τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, υπάρχει μία συμμετοχή σε μία συμφωνία προαιρετικά. Για όλα τα υπόλοιπα θα συνεργαστώ με μεγάλη χαρά με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω να μπορέσω να συμμετέχω κι εγώ σε έναν ε, καλό συμβιβασμό μεταξύ των διαφορετικών απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό αυτό το θέμα γιατί στο μέλλον ε, ενδεχομένως όλες ε, οι μελλοντικέ συμφωνίες ε, θα αναφέρονται στην ενεργειακή πολιτική, ειδικότερα για τις πρώτες ύλε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σεβαστό, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, να ξέρουμε ακριβώς τη σύνδεση της ενεργειακής πτυχής με την συμφωνία. Γι' αυτό υποστηρίζω την προσέγγιση αυτή του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής μας, ώστε να είμαστε βέβαιοι στο μέλλον ε, ότι ε, σε συμφωνίες όπως η ΣΥΤΑ, η TTIP, κάθε φορά που συζητούμε για ενεργειακές ε, πολιτικές, να υπάρχει συνεννόηση σε επίπεδο κρατών μελών. Κάτι ακόμη το θέμα της επικουρικότητας. Αν υπάρχει μια διεθνής ε, συμφωνία για την ευθύνη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για την ενεργειακή πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη ανταλλαγή απόψεων και να λαμβάνονται υπόψη ε, οι απόψεις και τα δημοκρατικά δικαιώματα του περιφερειακού επίπεδου, ποιες ε, είναι η, ποια θα είναι δηλαδή η συμμετοχή των ε, δήμων και κοινοτήτων ε, στην ενεργειακή πολιτική, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διαμόρφωση των διεθνών συνθήκων. Οπότε... Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεργαστούμε στενά με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ομάδα μου. Είναι πολύ σημαντικό οι συμφωνίες μεταξύ κρατών ε, στο τομέα της ενέργειας να συμφωνούν με το δίκαιό μας και με τους στόχους μας. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Σόλτς. Χαιρετίζουμε λοιπόν την τροπολογία 4 του συναδέλφου Μπένσεν που αναφέρεται στη στρατηγική της Ένωσης. Φυσικά στηρίζουμε και τις τροπολογίες 5 και 6 που σχετίζονται με το εμπόριο. Ένα πρόβλημα που ήδη αναφέρθηκε είναι τι γίνεται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνάπτουν συμφωνίες. Γιατί συχνά έχουμε μια δυσχέρεια. Κάτι παρουσιάζεται ως ε, ιδιωτική, ως ιδιωτική επιχείρηση αλλά το κράτος ε, είτε παίζει ουσιώδη ρόλο είτε έχει και την ε, πλειονότητα των μετοχών. Πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε αυτό και αναφέρομαι στην τροπολογία 2 που το αντιμετωπίζει. Γιατί το θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι αρκετά λεπτό. Σε αυτή τη συγκύρια Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το τι πρέπει να κάνει και τι όχι η Ένωση στα κράτη-μέλη. Δηλαδή πώς εφαρμόζεται η επικουρικότητα. Είναι λοιπόν πολύ λεπτό αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά πρέπει παρόλα αυτά να το λάβουμε υπόψη. Χαίρομαι γιατί ε, προβλέπω ότι θα έχουμε πολύ επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είμα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Επιτροπή. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστή η εκ των πρώτων αξιολόγηση τη συμφωνία, τη υπογραφής συμφωνία μιας χώρας μέλου με τρίτη χώρα. Αλλά θεωρούμε όχι μόνο στον τομέα του φυσικού αερίου, αλλά σε όλους του ενεργειακού τομεί. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους περιοριζόμαστε μόνο στον τομέα του φυσικού αερίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα συμφωνούσα με αυτό το ερώτημα. Μπορεί η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας να μας απαντήσει. Καλημέρα σα, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο, τον εισηγητή, του κοιόδης εισηγητές και τα μέλη τη Επιτροπής αυτή για το ενδιαφέρον του ω προ το θέμα αυτό και την υποστήριξη τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση είναι ένα σημαντικό τμήμα της Ενεργειακής Ένωσης, ώστε να υπάρχει συνοχή ε, στο, ενεργειακό κομμάτι στο κομμάτι της ενεργειακής πολιτικής ε, και συμφωνούμε επίσης ε, ότι η συνοχή και η συμβατότητα των συμφωνιών αυτών ε, με την ενωσιακή νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική για την οικοδόμηση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς. Σημειώσαμε τα ερωτήματά σας σε σχέση με το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις εμπορικές συμβάσεις που έχουν να κάνουν με τις συμφωνίες αυτές. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και εσωτερικά. Πρέπει να δούμε και τη νομική βάση και τι μας επιτρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο ε, των ε, συμφωνιών αυτών, δηλαδή το άρθρο 914 της ε, συνθήκης, μας θέσατε το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Εμείς έχουμε σκοπό να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ε, ε, Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει απόφαση στο πλαίσιο του Σώματος των Επιτρόπων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό για την αξιολόγηση. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ την Επιτροπή σας για την ε, υποστήριξή σας και ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε άλλα ζητήματα. Μήπως μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα για το θέμα των διαφόρων ειδών ενέργειας, γιατί συγκεκριμένα το αέριο, τι γίνεται με το πετρέλαιο και άλλες, ε, άλλους ενεργειακούς πόρους. Ναι, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα είδατε ότι όλα τα είδη καλύπτονται. Ε, η πυρηνική ενέργεια είναι τμήμα, ε, διέπεται από τη συνθήκη Ευρατόμ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καλύπτουμε το αέριο λόγω των προβλημάτων που είχαμε με κάποιες ε, συμφωνίες που είχαν επικεντρωθεί στον τομέα του αερίου. Αλλά είχαμε ζητήματα και με συμφωνίες που είχαν να κάνουν με το πετρέλαιο. Είναι και το πετρέλαιο σημαντικό. Είναι ένας σημαντικός υποψήφιος για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και για τον ηλεκτρισμό. Είναι επίσης σημαντικό να δούμε ότι στο μέλλον μπορεί να έχουμε σημαντικά έργα υποδομών, τα οποία θα χρειαστούν τέτοιου είδους συμφωνίες, οπότε κάποια στιγμή ε, πρέπει όλα τα είδη ε, της ενέργειας να καλύπτονται από την εκ των προτέρων αξιολόγηση. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο και πάλι στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπέντσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους σκιώδες εισηγητές για τα καλά του σχόλια και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είναι καλές οι διαπραγματεύσεις για να είναι και καλό το αποτέλεσμα για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και εγώ ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες ε, είναι 15 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας. Πάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση αυτού. Έχω το εξής πρόβλημα. Δεν είναι εδώ η συγητής μας. Κύριε Σόλτς, μπορείτε να τον αντικαταστήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής ε, ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να σας μεταφέρω το μήνυμά του, οπότε θα διαβάσω το έγγραφο των παρατηρήσεών του των εισαγωγικών για το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότηση Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευσή του. Ξέρουμε όλοι ότι το αέριο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπου το 1 τέταρτο τη ενεργειακή κατανάλωση και θα εξακολουθήσει να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του ενεργειακού μείγματο για, για, για, για το παρόν και το μέλλον. Η ενεργειακή ζήτηση και η ζήτηση αερίου θα αυξηθεί, δεδομένου ότι αυξάνεται και ο πληθυσμός. Αυτή τη στιγμή ε, θα, είναι, υπάρχει μόνο, θα είναι ε, μόνο το 10% των εισαγωγών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι ένα βασικό αγαθό και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανεξάρτητη από τους προμηθευτές αερίου, όχι μόνο για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και για να είναι ανταγωνιστική και συνεπώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαφοροποιημένων πηγών ε, προμήθειας. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο μπορεί να είναι εναλλακτικό καύσιμο και μπορεί να αντικαταστήσει τα ε, παραδοσιακά καύσιμα ε, και τη βελτίωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την ε, ε, μεταφορά του σε ε, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ πιο καθαρό σε σχέση με το ντίζελ, το αργό πετρέλαιο και άλλα είδη ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί πιο εύκολα να ε, μεταφερθεί και να αποθηκευτεί. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας και είναι πολύ σημαντικό στη σύναψη συμφωνιών όπως η TTIP ε, ως προς το ενεργειακό κεφάλαιο των συμφωνιών αυτών. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου που είναι μια βιώσιμη λύση για να υπάρχει μια οικονομία χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα. Για να υπάρχει υπάρχει όμως ε, βιώσιμη παραγωγή ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου, αερίου και ε, μεταφορά του, πρέπει να βελτιώσουμε την αγορά και την πρόσβαση στην αγορά, πρέπει να σταματήσουμε την ενεργειακή απομόνωση και αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και στο πλαίσιο του εμπορίου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου ασχολείται με αυτό το θέμα. Αναμένω σε συνεργασία με όλου του κοιόδη συζητητέ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σόλς. Θα να δώσω τώρα το λόγο σκιώδης εισηγητές. Ο κύριος Κέλλη δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος εδώ από το ΕΛΚ για να τον αντικαταστήσει. Εντάξει, τότε οι σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος Μαυρίδης. Να ευχαριστήσω τον ε, αντικαταστάτη του εισηγητή και τον εισηγητή και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης είναι μια καλή αφετηρία για τη συζήτησή μας σε αυτή τη φάση. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά. Πρώτον, η ανάγκη εξασφάλισης ε, ίσης πρόσβασης ε, σε ε, ενέργεια καλής, σε καλές τιμές. Το ε, γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος ε, εισαγωγέας ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο και συνεπώς αυτό δείχνει πόσο επίγονη είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προσπαθήσει να αναπτύξει τις δικές της ε, φυσικές, ε, τους δικούς τους φυσικούς πόρους, όπως για παράδειγμα τα κοιτάσματα που υπάρχουν στα ανοιχτά της Κύπρου, όπως επίσης και τη βελτίωση και τη δημιουργία ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Μεσόγειο θάλασσα, επίσης να εκμεταλλευτεί κοιτάσματα από την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, που είναι γειτονικέ περιοχές. Αυτό θα προωθήσει επίσης ε, το εμπόριο ως προς την ανάπτυξη οικονομιών ε, ε, κλίμακα. Επίσης, ε, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και η αποθήκευσή του έχουν μεγάλη σημασία για την αποφυγή τη εξάρτηση από έναν ενεργειακό προμηθευτή και ε, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ενεργειακή διαφοροποίηση και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ενεργειακή μα ασφάλεια. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε το φυσικό αέριο, το, να, υπάρχει, να υπάρχουν σταθμοί αποθήκευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βαλτική θάλασσα και στη Μεσόγειο. Τέταρτο σημείο, να τονίσουμε το γεγονός ε, ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο και η αποθήκευσή του είναι ένα σημαντικό τμήμα τη ενεργειακής πολιτικής τη Ευρωπαϊκής Ένωση και πρέπει να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή απομόνωση οποιαδήποτε κράτου μέλους ή περιφέρειε Ευρωπαϊκής Ένωση Και πέμπτον, η ανάγκη υποστήριξη των πιο ευάλωτων χωρών ε, στην προσπάθειά τους διαφοροποίησης των ενεργειακών ε, πηγών τους, ε, η σημασία του να υπάρξει αποτελεσματική από απόψεως κόστους ενέργεια, μακροχρόνια ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια για τις λιγότερο συνδεδεμένες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της και τα διεθνή φόρα για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ένα, μια ελεύθερη και διαφανής ενεργειακή αγορά σε όλο το κόσμο. Πρέπει επίσης να είμαστε πιο ε, προδραστική ε, όσον αφορά την εκστρατεία ε, για τα ενεργειακά δικαιώματα, τη σημασία τους στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες που εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο σέβονται τα απαραίτητα περιβαλλοντικά, τις απαραίτητες περιβαλλοντικές προδιαγραφές όπως επίσης και τους κανονισμούς ασφαλείας. Για το ECR τώρα, κ. Σαβαλή. Σαχαντήλ, συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ. ένα θέμα γεωπολιτικής φύσης αυτό. Το ξέρουμε όλοι. Και υπάρχουν χώρες στην Ένωση, Βαλτική και την Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ανατολική Ευρώπη, που εξαρτώνται αποκλειστικά από έναν προμηθευτή μόνο. Οπότε είναι ευάλωτες στην διακοπή της παροχής. Οπότε πρέπει να αναπτύξουμε τη δυνατότητα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές. Οπότε εδώ το ΙΦΑ μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Αυτό είναι το κυριότερο. Γι' αυτό η μέσο μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης θα πρέπει να διευκολύνει αυτή ακριβώς την πρόσβαση διαφοροποιημένη πηγέ προμήθειας και να αποφύγει ακριβώ την εξάρτηση από ένα μόνο προμηθευτή ή ένα μόνο σημείο διέλευση, Επειδή αυτό επιτρέπει βεβαίω καταχρήσει και κατάχρηση δεσπόουσας θέση και χειραγώγηση. Δεύτερον, ξέρουμε όλοι ότι και επιχειρήσεις αλλά και τα σπίτια στην Ένωση θα συνεχίζουν να εξαρτώνται στο άμεσο μέλλον από το φυσικό αέριο το υγροποιημένο. Ανεξάρτητα από την προσπάθεια μείωση παρουσία του άνθρακα στην αγορά ενέργεια στην Ένωση, κάτι το οποίο μακροχρόνιο μα στόχο. Λαμβάνοντα λοιπόν αυτό υπόψη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ εμπορίου και ενεργειακών πολιτικών σε σημαντικές περιοχές του κόσμου, Βορειοαφρική, Ασία, Αμερική και μάλιστα σε περιοχές όπου το εμπόριο ενέργεια δεν ρυθμίζεται σε πολυμερές επίπεδο. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να είναι και ο απότερος στόχος της Ένωσης, η δημιουργία δηλαδή ενό πλαισίου που θα μπορεί να διαχειρίζεται την ενέργεια, τα ενεργειακά προϊόντα και αυτό ας ελπίσουμε από την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Αυτά προς τον παρόν πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω και πρόεδρο. Ο κύριος Μπούχνερ τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα και την ομάδα μου είναι σημαντικό να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύνδεση με τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Οποιαδήποτε δηλαδή αύξηση της χρήσης τους. Γι' αυτό Πρέπει να δούμε με σκεπτικισμό οποιαδήποτε ενέργεια αυξάνει την χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτό το αναφέρει και ο συγκεκριτής του 6 και στο 7. Ιδιαίτερα η Κομισιόν τα τελευταία χρόνια έχει υπερεκτιμήσει κατά πολύ τις ανάγκες σε φυσικό αέριο. Και αυτό το επέκρινε και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης και της πολιτικής για το κλίμα μέχρι το 2030 θα πρέπει να ε, μειώσουμε ακόμη περισσότερο τις προβλέψεις χρήσης φυσικού αερίου. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 6. Κάτι άλλο. Η έκθεση θεωρεί ότι θα υπάρξει μείωση του υγροποιημένου αερίου σε σχέση με το αέριο που περνάει μέσω από αγωγούς. Αυτό θεωρώ ότι είναι αμφίβολο, γιατί υπάρχουν πολύ ουσιώδεις διαφορές από πλευράς τεχνολογίας. Πάντα θα υπάρχει διαφορά στην τιμή. Ο τρόπος για να μειωθεί αυτή η διαφορά στην τιμή θα έπρεπε να περνάει, για παράδειγμα, να, περάσουμε μέσα από το TTIP για να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την υδρορογμάτωση, το fracking. Αλλά αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Επίσης, στην παράγραφο 4 αναφέρονται οι προδιαγραφές για την εξόριξη του φυσικού αερίου και λέγεται ότι πρέπει να τηρούνται οι δικές μας ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεν πρέπει να εισάγουμε φυσικό αέριο το οποίο εξορίσεται μέσω fracking με μεθόδους δηλαδή που δεν επιτρέπονται σε μας. Γι' αυτό θέλω να τονίσω συγκεκριμένα ότι ναι μεν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το fracking, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι δικές μας προδιαγραφές και κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι εδώ ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικέ λύσεις. Ο κλάδος, από ό,τι φαίνεται, προσανατολίζεται προς αντιμετώπιση της ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο με ένα τρόπο που τον αναφέρει ως τεχνητό φυσικό αέριο. Δηλαδή να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν εδώ και χρόνια για να παράγουμε αέριο. Για να τροποποιήσουμε μάλλον το αέριο. Αυτή η εξέλιξη οπωσδήποτε θα επηρεάσει πολύ και τις εισαγωγές μας. Γι' αυτό θέλω και αυτή η ε, αντιμετώπιση να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπορέλη και μετά θα πάρει το λόγο και ο κύριος Κέλλη. Αλλά πρώτα ο κύριος Μπορέλη και μετά εσείς. Ευχαριστώ πολύ και εγώ στο συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λόγω της σημασία του ζητήματος και του γεωπολιτικού πλαισίου, νομίζω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να προχωρήσει πιο μακριά από την απλή ανταλλαγή απόψεων. Να αναφέρω κάποιες σκέψεις που μετά θα αναπτύξω υπομορφή τροπολογιών για να συμβάλλω σε αυτό το φάκελο που νομίζω ότι έχει εξεταστεί εντελεχώς και στην ίντρη στην οποία ανήκω. Ως γενική αρχή η ενέργεια είναι ένας βασικός παράγοντας της αναπτυξής μας. Σήμερα όμως διδραματίζει ένα κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Κυρίως λόγω της, ε, των δυσκολιών, των ισχυριών που αντιμετωπίζουμε στη γειτονιά μας παλαιότερα υπήρξε σταθερότητα, σήμερα όχι. Αυτή λοιπόν η αστάθεια σήμερα έχει επιπτώσει και στην ενεργειακή προμήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω εξάλλου έχει σημειώσει και η Κομισιόν. Στο σημείο 2, σύμφωνα με αυτά που είπε η Κομισιόν, θα πρέπει να διερευνήσουμε νέε εταιρικέ σχέσει στον τομέα τη ενέργεια, να απαλυθεύσουμε τι υπάρχουσε και με τους τωρινούς εταίρους να αναπτύξουμε ένα διάλογο με ad hoc εταιρικές σχέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ωφέλιμες. Για το σημείο 3 συμφωνώ για τους στόχους τους ευρωπαϊκούς όσον αφορά το περιβάλλον και την ε, αλλαγή του κλίματος. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στην ενεργειακή απόδοση. Ένας, ε, σημαντικής, ένας σημαντικός τομέας για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από διάφορους προμηθευτές και ταυτόχρονα να βλιστοποιήσουμε την κατανάλωση. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται μόνο με το διεθνές εμπόριο, αλλά είναι σαφές ότι μια πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας έχει άμεσες επιπτώσεις στις ανάγκες μας και κατά συνέπεια στις εμπορικές μας σχέσεις που θα συναυθούν. Όπως επαναλαμβάνει συχνά το έγγραφο της Κομισιόν, έμεσα αναφέρεται στο 4 εξάλλου, ένα βασικό ζήτημα είναι το θέμα των υποδομών. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία τους, αλλά ειλικρινά το να δώσουμε έμφαση στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής είναι μια προοπτική η οποία μας ανησυχεί. Θα προτιμούσαμε αντίθετα να αναθεωρήσουμε τις τωρινές δυνατότητες, να αξιολογήσουμε καλύτερα τη χρήση των τωρινών υποδομών σε όλα τα επίπεδα, αγωγούς, αποθήκευση, διανομή και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των τωρινών υποδομών παρά να χτίσουμε νέες. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τις ε, επιπτώσεις και στις τωρινές κοινότητες αυτών των υποδομών και την συμμετοχή των κοινότητων αυτών στην εργασία λήψη αποφάσεων. Η αγορά είναι υπερβολικά αισιόδοξη καμιά φορά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό αριθμό υποδομών σε σχέση με, με επίπεδα κατανάλωσης που δεν απαιτούν τέτοιες εγκαταστάσεις. Επίσης, ε, σημαντικό θεωρώ είναι, ότι είναι να υπάρχει διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις της διεθνής όσον αφορά την ενέργεια. Και τέλος, όπως αναφέραμε στο 5, η ανάγκη εξέλιξης και μετάβασης σε μια χαμηλότερη παρουσία του άνθρακα στον τομέα της ενέργειας μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή για Ευχαριστώ. Να και εγώ να στήσω συγγνώμη. Είχα ψηφοφόρους το πρωί. Καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης ώστε να έχουμε μια τελική άποψη στους επόμενους δύο μήνες. Εξελίσσεται ταχαία η αγορά φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα για την Ευρώπη δύο σημαντικά ζητήματα. Ενεργειακή ασφάλεια και εξέλιξη των τιμών. Η διεθνή μας λοιπόν στρατηγική είναι κεφαλαίου σημασία και συμφωνώ με τι απόψει του εισηγητή για την ενεργειακή ασφάλεια. Καλωσορίζω και την ανακοίνωση τη Κομισιόν για νέα στρατηγική για το ΙΦΑ και την αποθήκευσή του και τι ευκαιρίε που παρουσιάζει για την ενεργειακή ασφάλεια. Η ενεργειακή αγορά και η παρέμβασή μα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο Αντιμετώπιση του μοναδικού προμηθευτή και την ενίσχυση της ηθαγενή παραγωγής στην Ευρώπη. 119 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα είχαμε το 2015 στην Ευρώπη, 14% λιγότερα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε εισαγωγές. Το 2015, 41% λοιπόν των εισαγωγών μας φυσικού αερίου ερχόταν από τη Ρωσία. και είχαμε περισσότερο το 15 από το 14 παρά τις κυρώσεις λόγω της παρεμβάσης στην Κρυμαία. Θα πρέπει λοιπόν να απομακρυνθούμε από αυτή την εξάρτηση ανεξάρτητα από την άποψη που έχουμε για την Ρωσία ως μοναδικό προμηθευτή. Είναι κακό αυτό για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και στην ουσία θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τους αγωγούς που αφορούν μόνο τη Ρωσία και να χτίσουμε νέους. Αν δούμε Άλλε χώρε θα δούμε τι έγιναν, τι προσπάθειες έγιναν για τη μείωση αυτή της αποκλειστική προμήθειας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφοροποίηση αναχώρα, θα πρέπει να αναπτύξουμε 4,9 δις τετραγωνικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ζήτηση, μειώνοντα τι ρωσικέ εισαγωγέ. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη όπου οι δράσει αυτέ ε, ήταν, ήταν αποτελεσματικέ. Πάνω χάρη η χώρα μου, η Ιρλανδία, από το Δεκέμβριο του 2015 εξαρτώμασταν από έναν αγωγό από το Ηνωμένο Βασίλειο για το 95% του αερίου που ερχόταν στη χώρα μας. Είχαμε νέα κοιτάσματα στη χώρα μας που θα αποδώσουν το 2022 και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην ε, εξαρτώμαστε μόνο από μια χώρα της Ένωσης και οι επιπτώσεις του Brexit θα έχουν και αυτές μεγάλες επιπτώσεις. Μια σημαντική εξέλιξη στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας πρόσφατα είναι η σύγκληση τιμών στην Ασία και στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να το υποτιμήσουμε γιατί θα δημιουργηθεί μια παγκόσμια αγορά και ο ανταγωνισμός θα, έχει, οδηγήσει στην πίεση των τιμών. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν, ε- Ένωση θα μπορούσε να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τη, επωφελούμενη από αυτή την κατάσταση. Η αποθήκευση του ΙΦΑ θα πρέπει να οδηγήσει στην βελτίωση τη απόδοση, της απόδοσης και στην διαφοροποίηση τη προμήθεια. Οι ΑΠΕ από τους δεν επαρκούν και το φυσικό αέριο μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά, ενεργειακά συστήματα μέσω πρόθεσμα. Γι' αυτό ακριβώ αυτή η στρατηγική θεωρώ ότι είναι έγκαιρη και κέρια. Θα πρέπει να καλύψουμε βεβαίω τα κενά μακροπρόθεσμα για τις ΑΠΕ και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τι προκλήσει για το περιβάλλον, δημιουργώντα ένα νέο ενεργειακό σύστημα. Αλλά αυτό δεν θα γίνει από μια νύχτα στην άλλη. Η ισορροπία λοιπόν μεταξύ αερίου και ΑΠΕ θα πρέπει να μα οδηγήσει στην μείωση τη χρήση του άνθρακα και να σα πω επίση ότι το 2015 είχαμε χαμηλέ τιμές στο φυσικό αέριο, κατά το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ θετική εξέλιξη. Και καλωσορίζω την έκκληση του εισηγητή να υπάρχουν ενεργειακά κεφάλαια στι ναι, εμπορικέ συμφωνίε τη Ένωση. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό και η TTIP εδώ είναι ένα σημαντικό παράδειγμα. Η δυνατότητα εξογής 12,2 δισεκατομμύρια τετραγωνικών μέτρων προήρθε από το Τέξας και μόνο και από την δημιουργία υποδομής στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. Και έχουμε νέα κοιτάσματα με 17 δις τετραγωνικών μέτρων φυσικού αερίου. Αυτή η επιπλέον ποσότητα θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές του αερίου στην Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώ τα πλαίσια της TTIP αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητά μα. Τέλο, η αποτελεσματική χρήση των υποδομών είναι πολύ σημαντική θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν και νέα προγράμματα αγωγών το ταχύτερο δυνατόν με σύνδεση και τέρμιναλ ώστε να έχουμε ένα, μια ενιαία αγορά φυσικής, φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πολλά από αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να συνοδεύονται από, τη, αποφάσεις για τις επενδύσεις και θα πρέπει να γίνει αυτό το ταχύτερο δυνατό για να ωφελήσει το σύνολο της Ένωσης. Καταλήγοντας, χαιρε, ε, συγχαίρω τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του και προσβλέπω στη συνεργασία με εσά και τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριο Σόλτστορ. Ευχαριστώ. Να αναφερθώ σε δύο θέματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, ε, η γεωπολιτική πλευρά. Πολλά μπορούμε να πούμε για την εξάρτηση από συγκεκριμένους ε, εισαγωγείς ε, τους Ρώσους και πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας. Όμω πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί. Όταν συζητάμε για τα εμπορικά θέματα, πρέπει να συζητήσουμε και τιμέ. Και για τη διαμόρφωση των τιμών πρέπει να λάβουμε στο μέλλον πολύ περισσότερο. Ε, να λάβουμε λοιπόν υπόψη πολύ περισσότερο διάφορους παράγοντες όπως η οικολογική παραγωγή και η μεταφορά. Μόνο έτσι θα έχουμε μια σωστή, μια ε, έντιμη σύγκριση των τιμών Χρειαζόμαστε βεβαίως περισσότερες ανανεώσιμες. Αλλά υπάρχουν μελέτες της Κομισιόν που αναφέρονται στους τερματικούς σταθμούς για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Και λένε ότι όταν μιλάμε για τα κρουαζιερόπλια στα λιμάνια, υπάρχει μια πηγή, ή μάλλον θέλουμε, να οικοδομήσουμε τροφοδοσία σε ηλεκτρικό, που θα είναι πιο φτηνή από τη χρήση φυσικού αερίου. Θα είναι πιο φτηνό έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα από το ρεύμα που παράγουν τα ίδια τα πλοία στα λιμάνια. Άρα θα είναι πιο καθαρή αυτή η πηγή ενέργειας και θα μολύνει περισσότερο τα λιμάνια και άρα θα επιβαρύνει, θα μολύνει λιγότερο, συγγνώμη, τα λιμάνια και άρα θα επιβαρύνει λιγότερο και τους κατοίκους των λιμανιών. Στην δική μου εκλογική περιφέρεια υπάρχει πολύ έντονη ζήτηση γι' αυτό. Πρέπει στα λιμάνια να χτίσουμε σταθμούς χρήσης LNG που θα παράγουν ρεύμα για τα κρουαζιερόπλια ή θα συνδέσουμε τα κρουαζιερόπλια απευθείας με το ηλεκτρικό ρεύμα το γενικό της περιοχής. Άρα σε τι βαθμό θα βοηθήσουμε τις περιφερειακές πηγές παραμονής ενέργειας. Στο Αμβούργο για παράδειγμα χτίστηκαν τέτοιοι σταθμοί ε, χρήσης LNG στο Ρόστοκ όμως προτίμησαν ε, το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο παράγεται γενικά, γιατί μακροπρόθεσμα είναι πιο ασφαλής πηγή και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Και άρα σε τελευταία ανάλυση και καλύτερη τιμή, αλλά επιτυχάνουμε έτσι. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Αλλά οι μεγάλες εταιρείες μα ε, μας λένε όχι, έχουμε καλύτερα φίλτρα για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για τα καύσιμα, έτσι έχουμε τη δική μας ε, προμήθεια σε ενέργεια και προβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα. Θέλω λοιπόν να πω ότι, όταν συζητάμε τέτοιες γνωμοδοτήσεις ως Επιτροπή πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τέτοια πολύ πρακτικά θέματα για τις τοπικές αρχές, για την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Αυτός πρέπει να είναι πάντα ο κύριος στόχος μας. Να έχουμε ασφαλή ενέργεια με βάση τις τοπικές πηγές και με σωστή πρόβλεψη για το πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες μας ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα, η ΕΜΑ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, συμφωνούμε όλοι ότι η Ένωση πρέπει να έχει ένα ενεργειακό μοντέλο όπου έχουν σημαντική παρουσία οι ΑΠΕ και να μην έχουμε την εξάρτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή για τις βασικές μορφές ενέργειας. Θεωρώ λοιπόν ότι όντως αυτό που πρέπει να κάνουμε μια στρατηγική και αυτό διέρχεται βέβαια από τη διπλωματία, από συμφωνίες με τους μεγάλους προμηθευτές και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια καλή μελέτη για τις ανάγκες υποδομής όσον αφορά τη διανομή και την αποθήκευση για το ΙΦΑ. Εξάλλου νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό παρουσιάζεται ως χρήση του ΙΦΑ για τα πλοία. Και μάλιστα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα συγχρηματοδούμενο από την Ένωση όπου έχουμε μετατροπή ενός πλοίου υψηλής ταχύτητας για την χρήση του ΙΦΑ. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποια είναι η σχέση αυτή τη στιγμή που έχουμε μεταξύ όλων αυτών των στοιχείων ώστε να έχουμε καλές προοπτικές για τη χρήση του υγροποιημένου ως και ενεργητική, ενεργειακή πηγή αλλά και ως ε, πηγή καυσίμου για τις μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yes, uh, thank you very much. This was really... Ευχαριστώ. πολύ σημαντική συζήτηση για μας για να λάβουμε υπόψη στις περαιτέρω ενεργές μας. Το LNG θα βοηθήσει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια προμήθειας, την ασφάλεια φοδιασμού. Πρώτα απ' όλα θέλουμε περισσότερη διαφοροποίηση. Ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες περιοχές, όπως η Ανατολική Ευρώπη, η Βαλτική, και η Βυρική Χερσόνησος. Και όπως υπόθηκε, τρεις άξονες έχουμε. Πρώτον, να ολοκληρώσουμε την αγορά με την αναγκαία υποδομή και συμφωνούμε ότι πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η υπάρχουσα υποδομή και προσεκτικά να επιλέξουμε τι πρέπει να προσθέσουμε επιλέγοντας ε, τις πιο χρήσιμες ε, τις πιο βιώσιμες. Για την αποθήκευση τώρα. Πρέπει να υπάρχουν ε, συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού για την αποθήκευση. Δεν υπόθηκαν πολλά για την αποθήκευση, αλλά είναι βασική για την ασφάλεια εφοδιασμού. Γιατί αν υπάρξει μια διακοπή της παροχής, πρέπει να έχουμε αποθηκευμένες ποσότητες. Και βεβαίως Πρέπει να υπάρχουν διαφανείς τοπικές αγορές μέσω πολυμερούς και διμερούς διαλόγου. Έχουμε και σημαντικούς ε, στόχους για την κλιματική αλλαγή και θέλουμε οπωσδήποτε να επιτύχουμε τους στόχους ε, της διάσκεψης των Παρισίων, να αυξηθεί η χρήση ανανεωσίμων. Το φυσικό αέριο και το LNG ε, θεωρούμε ότι είναι απλώς μεταβατικές πηγές που θα μας χρησιμεύσουν μέχρι να εισαγάγουμε στο μείγμα πολύ περισσότερες ανανεώσιμες. Υπόθηκαν πολλά για τις προβλέψεις ε, ζήτησης ε, φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αναμένουμε μία μικρή μείωση της κατανάλωσης αερίου τα επόμενα χρόνια και η ενδογενής παραγωγή επίσης μειώνεται, αυτό σημαίνει ότι οι εισαγωγές θα παραμείνουν σταθερές πάνω κάτω. Γι' αυτό χρειαζόμαστε διαφοροποίηση, για να υπάρξει περισσότερη απεξάρτηση. Και τέλος, το LNG συνδέει τις υπήρους και επειδή ε, είναι προϊόν αγοραπολισιών παντού στον κόσμο, ότι γίνεται σε μια περιοχή, επηρεάζει τις άλλες μόνο μια ρέουσα και διαφανής αγορά θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τους κραδασμούς και τις διακοπές. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε διάλογο με τους εταίρους μας παγκοσμίω και με τους καταναλωτές και τους παραγωγούς και θα εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, αλλά επίση και με τον Καναδά και την Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ο Χέλμουτ από πλευράς ε, του εισηγητή ο κύριος Σόλτς. Ναι, ο εισηγητής ε, μου ζήτησε να ευχαριστήσω τους Κιώδης, όλους τους άλλους που πήραν το λόγο για την συμβολή τους τον εμπλουτισμό της εργασίας, του σχεδίου, του κειμένου του. Οπότε θα επανέλθει με περαιτέρω προτάσεις για την περαιτέρω επεξεργασία αυτού του σημαντικού θέματος. Θα είναι σε επαφή συνεχώς με τους κοιόδης και ελπίζει ότι θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, προθεσμία για τροπολογίες 15 Ιουλίου 18. Η ψηφοφορία θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου. Και τώρα να περάσουμε στο 8, και αυτό πολύ σημαντικό, Γενικός Προπολογισμός της Ένωσης για τον επόμενο χρόνο. Όπως θα θυμάστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο με κάποια καθυστέρηση φέτος. Μετά από τη θαυμαστή πέμπτη για την Βρετανία, την υπέβαλε λοιπόν στις 30 Ιουνίου, άρα οι προθεσμίες ε, είναι πολύ σφιχτές αλλά το θέμα είναι προφανώς σημαντικό ιδιαίτερα για το εμπόριο. Πρέπει να στηρίξουμε τον προπολογισμό του εμπορίου, γιατί το εμπόριο είναι η κινητήρια δύναμη του βιωσίμου ε, Συγγνώμη, ναι, το εμπόριο είναι η κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη και δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό η πρόταση της Κομισιόν, αλλά να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέγκε, που είναι ο ειδικό μας ως εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πολύ καλά νέα είναι βέβαια ότι όλη η συζήτηση για το πώς θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 της συνθήκης και το τι είδους ε, συμφωνίες θα πρέπει να διαπραγματευτούμε δεν είναι τμήμα το, της συζήτησης για τον προϋπολογισμό για το 2017. Βέβαια κανένα, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τώρα ε, τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την, ε, τη συζήτηση για την αναθεώρηση του ε, ευρύτερου πλαισίου του προϋπολογισμού. Είναι μια πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα πλέον, αλλά δεν είναι ε, τμήμα της τωρινής μας εργασίας. Αναφερθήκατε στο ότι υπήρξε μια καθυστέρηση και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Έχουμε τώρα προγραμματίσει ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότησης θα είναι η 18η Ιουλίου για δημοσιονομικές τροπολογίες συγκεκριμένες δημοσιονομικές θέσεις 3 Αυγούστου και Νομίζω ότι έχουμε προγραμματίσει 31 Αυγούστου την ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ο Γενικός Τριμερής Διάλογος μεταξύ των ε, θεσμών θα λάβει χώρα Σεπτεμβρίου. Και ε, επειδή ακριβώς έπρεπε να κάνω μία σύνοψη της, ε, του σχεδίου γνωμοδότησης πριν από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, είχα ακόμη κάποιες ε, ιδέες που έχουν συμπεριληφθεί στο έγγραφο που είναι διαθέσιμο στο φάκελό σα, Για παράδειγμα, δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ιδέα ενό προγράμματο Juncker 2 για την Αφρική. Τι σημαίνει αυτό, τι αντίκτυπο έχει κάτι τέτοιο, για παράδειγμα για τον προπολογισμό, τι σημαίνει για τι ε, δραστηριότητε μα ω επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και επίση πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις εξελίξεις, γιατί ένα από τα ευαίσθητα θέματα είναι ότι λόγω της διαχείρισης κρίσεων και της κινητοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων ε, και των ε, μέσων ε, ευελιξίας που τις χρειαζόμαστε απελπισμένα κατά την περίοδο κρίσης είναι σημαντικό να έχουμε έναν προπολογισμό για να ανταποκριθούμε στην κρίση, την προσφυγική. Από την άλλη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τέλος, να μην έχουμε πρόβλημα με τις πληρωμέ μας και η ενότητα του προϋπολογισμού να μην υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Εδώ έχω ένα ε, δελτίο που δείχνει ακριβώς ε, ε, την ενότητα του προϋπολογισμού και βλέπουμε ότι ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι και αυτό αντικείμενο, αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελέγξουμε ε, καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και ο Γιάννη Γκάιερ το ανέφερε αυτό σε κάποια από τα προπαρασκευαστικά του έγγραφα για τον τριμερή διάλογο, ότι για παράδειγμα αυτά τα δύο ταμεία, το Μαντάντ και το Ταμείο για τη Βόρεια Αφρική, να πάρουμε κάποια χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από τα υπάρχοντα προγράμματα γειτονίας και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη προαιρετικές εισφορές. Ε, αυτή τη στιγμή 69 εκατομμύρια είναι οι εθνικές εισφορές στο ΜΑΤΑΔ και 88 εκατομμύρια στο Ταμείο για τη Βόρεια Αφρική ήταν 500 και 150 ε, στο παρελθόν όμως πληρώνεται ένα ελάχιστο στην Διευθύνουσα Επιτροπή για να διατηρηθούν ε, οι ελάχιστες εισφορές των κρατών μελών. Αυτή δεν είναι όμως ε, μία μέθοδος που μπορεί να μας επιτρέψει να οργανώνουμε τις δραστηριότητές μας και τον προϋπολογισμό μας στο μέλλον, γιατί φαίνεται ότι με τέτοιου είδους εισφορές ε, τα ποσά τα οποία έχουμε προγραμματίσει και τα οποία αναμένουμε δεν θα έρθουν και από την άλλη αυτή η εξέλιξη δεν συνάδει με την ενότητα του προϋπολογισμού. Τώρα, για κάποια συγκεκριμένα σημεία είναι ε, προφανώς ε, σαφέστατο ότι η πρόταση του προϋπολογισμού για το 2017 ε, έχουν κάποιες κατηγορίες που είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντας να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή κάθε δυνατή ευελιξία για την προσφυγική κρίση. Αυτό βέβαια πρέπει να υποστηριχθεί. Από την άλλη όμως πρέπει να επιμείνουμε ότι θα υπάρξουν πιστώσεις υποχρεώσεων ε, στις εμπορικές δημοσιονομικές γραμμές ε, και ότι ε, πρέπει να γίνουν σεβαστές, να υπάρχουν δηλαδή τα απαραίτητα οικονομικά μέσα να αντιμετωπιστεί η κρίση των μεταναστών προοδευτικά σε διεθνές επίπεδο νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη θέση και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ε, ε, τόπων συγκέντρωσης των, ε, ε προσφυγών, των προσφύγων. Ε, ελπίζουμε να μην ε, βγούμε εκτός πορείας και να μην χρειαστεί να ξαναδούμε αυτές τις εικόνες που είδαμε πριν από μερικούς μήνες. Βεβαίως πρέπει να επιμείνουμε ε, να υπάρξει υποστήριξη στο εμπόριο και στις χώρες ανατολικής γειτονίας και τις χώρες αραβικής άνοιξης. Είναι κάτι το οποίο το έχω αναφέρει ήδη. Έχω αναφέρει το πρόβλημα των, χρηματοδοτικών μέσων εκτός ε, του προϋπολογισμού και η αξιολόγηση ε, της μη εξωτερικής ανάθεσης της αντιμετώπιση του προβλήματο αυτού πρέπει επίσης να υποστηριχθεί. Είναι σημαντική λοιπόν η ανταπόκρισή μας στην ε, αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων. Από την άλλη πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο έλιγμων για άλλα πολυετή προγράμματα η οποία μειώνεται βέβαια η δυνατότητά μας, η δυνατότητά μας αυτή κατά συνέπεια. Και θα σας πω κάποια ε, ποσά που θα μειωθούν πάρα πολύ όσον αφορά τις πληρωμές, ε, το μέσο ευρωπαϊκής ε, γειτονίας περίπου στο ίδιο επίπεδο, αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ε, στην, ε, στην Ε, στα, υπόλοιπα μέσα εκτός προϋπολογισμού της γειτονίας. Έχουμε ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη έρευνα για το πώς, μια ολόκληρη μελέτη για το πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα μέσα εταιρικών σχέσεων. Μήπως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει λίγο περισσότερες πληροφορίες. Πότε θα δημοσιευθεί αυτή η μελέτη. Νομίζω ότι είναι μελέτη της ΕΙΕΔ δεν έχει ακόμη πληρωθεί. Τι θα κάνουμε με τα νούμερα που βλέπουμε τώρα ε, στον προϋπολογισμό του 2017. Γνωρίζω επίσης ότι οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα πιλωτικά προγράμματα. Άκουσα τώρα ότι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις αναμένεται στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Και βεβαίως ε, αυτό μετά θα περάσει στα χέρια της Επιτροπής Προπολογισμού και των ε, αρμοδίων εισηγητών και σκιωδών εισηγητών για να δουν ποιες ε, θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας και να συμπεριληφθούν βεβαίως οι προτεραιότητες αυτές. Αυτά ήθελα να σας πω για την ώρα και ε, με χαρά θα περιμένω τα σχόλιά σας και ενδεχομένως τις ε, τροπολογίες σας επί του προπολογισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπέγκε. Να δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης συζητητές, ο κύριος Σούστα. Ευχαριστώ για την εισαγωγή του κύριο Μπέγκε και συμμερίζομαι τι απόψει του για πολλά σημεία. Συνολικά νομίζω ότι αυτός ο προπολογισμό είναι απόλυτα ανεπαρκής ε, έναντι των προκλήσεων που έχουν προκύψει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης ε, θα προκύψουν και άλλα λόγω του Brexit. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να έχουμε δυνατότητα να ε, αντιδράσουμε. Ωστόσο, ο προπολογισμό φυσικά είναι στα πλαίσια των πολιετών προοπτικών. Σε πολλούς τομείς λοιπόν Βεβαίως και πολλά θέματα ε, λοιπόν δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς ε, στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Πρέπει να τα συζητήσουμε από κοινού με άλλες επιτροπές. Και συνολικά το Κοινοβούλιο μόνο μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Οπότε για ένα θέμα θέλω να μιλήσω, όπου νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουμε έχουμε εισαγάγει διαδικασίες ελέγχου και αναμένουμε από την Κομισιόν αυτές οι διαδικασίες ελέγχου και επίβλεψης να χρηματοδοτούνται επαρκώς και εγκαίρως. Αυτό δεν έχει συμβεί πάντα στο παρελθόν. Νομίζω όμως ότι υπάρχει ετοιμότητα για να γίνει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήδη και σε αυτή την ε, συνεδρίαση αναφερθήκαμε σε εμπορικές συμφωνίες ε, που περιέχουν, που περιέχουν λεπτά σημεία και που πρέπει να μπορούν να επιτηρηθούν κατά την εφαρμογή τους. Αυτή η διαδικασία επίβλεψης, εποπτείας, πρέπει να συμπεριλάβει και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν ε, επαρκής βάση συμφωνίας για το θέμα αυτό, ότι θα καταλήξουμε σε συνενετικές διατυπώσεις. Θα μας ενδιέφερε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τις διαδικασίες αυτής, αυτές της εποπτείας και αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κέμπερ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε επιφυλακτικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που για πρώτη φορά εδώ και χρόνια αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Μας ανησυχούν οι πιστώσεις για το εμπόριο που είναι κάπως περιορισμένες, όπως είπε και ο συνάδελφός μου τώρα προηγουμένως. Και ο διαχωρισμός που γίνεται Οπότε οι ερωτήσεις. Γιατί μειώνται τόσο πολύ οι πιστώσεις για το MFA και η Γενική Διεύθυνση θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε επαρκές, προσωπικό επαρκής πόρους για όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουμε το TTIP και τώρα ακόμη έχουμε και την Βρετανία που θα προσθεθεί. Υπάρχει λοιπόν θέμα ανθρώπινου δυναμικού. Ε, ξέρετε ότι και η δική μας η πλευρά η Βρετανία ανησυχεί για το αν έχει το επαρκές και το κατάλληλο προσωπικό για τις διαπραγματεύσεις από πλευρά τη. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα και από τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ πολύ. Άλντε παρακαλώ. Η Μαρίτια νομίζω. Ποιος θα την αντικαταστήσει. Κανείς. Οκ. Okay. Και από τις άλλες ομάδες δεν βλέπω κανένα σκιώδη εδώ. Α, ο Χέλμουντ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που αναφέρθηκε στην περιπλοκότητα του θέματος στην εισαγωγική του παρουσίαση. Και σε άλλες εκθέσεις του κυρίου Μπέγκε έχουμε συζητήσει το θέμα της μακροπρόθεσμης ε, επάρκειας του προϋπολογισμού της Ένωσης. Και έχουμε πει ότι πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι εάν δεν αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης της Ένωσης, δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στα τόσο πολλά επιπλέον καθήκοντα και στις δραματικές εξελίξεις. Δηλαδή πρέπει να δούμε τους ίδιους πόρους. Πρέπει να δούμε με τι τρόπο θα πρέπει τα κράτη-μέλη με κοινοτικό πνεύμα να βοηθήσουν για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα να αναδιαμορφώσει τα έσοδά της. Γι' αυτό νομίζω ότι το 2 του σχεδίου του κύριου Μπέγκε είναι πολύ σημαντικό γιατί σημειώνει ότι το εμπόριο έχει να κάνει με την ανάπτυξη άλλων περιοχών του κόσμου. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα αίτια των μεταναστεύσεων, τότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις. Και ε, γι' αυτό παίζει ιδιαίτερο ρόλο το εμπόριο. Αυτό είναι ευρύτερο από το θέμα αυστηρά του προπολογισμού, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε στα πλαίσια της διαμόρφωσης του προπολογισμού. Επίσης, το θέμα των πόρων, των πιστώσεων δηλαδή, για το εμπόριο, και το κατά πόσο ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις τόσες συμφωνίες που έχουμε διμερείς, πολυμερείς κτλ. Και το τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε σε μερικά χρόνια. Και το θέμα των μικτών συμφωνιών. Όλα αυτά τα θέματα απασχολούν τους πολίτες. Πρέπει να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει, τι επιπτώσεις έχει για αυτούς η σύναψη συμφωνιών. Και επίσης για τη συμβολή των κρατών μελών. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια λοιπόν της πολιτικής εμπορίου για το πώς χρηματοδοτείται και πώς δαπανώνται οι πιστώσεις για το εμπόριο. Όσον αφορά τις εγγύσεις που δίδουμε εκτός Ένωσης, θα ήθελα ο συγητής να είναι πιο κατηγορηματικός. Δεν είναι δυνατόν ε, να αλλάζει ε, ο τρόπος χρήσης προγραμματισμένων πιστώσεων για να καλύψουμε κενά που προκύπτουν αλλού. Πρέπει να δράσουμε με υπεύθυνο τρόπο. Θέλω ο εισηγητής μας να είναι ιδιαίτερα άκαμπτος για τα θέματα αυτά και πρέπει να πει και στην Κομισιόν ότι το σχέδιο, προπολογισμό πρέπει, το σχέδιο προπολογισμού πρέπει να θέτει και το Συμβούλιο ενώπιον των ευθυνών του και σας ευχαριστώ. Ο Ντέιβιντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα για να συμφωνήσω με κάποια σημεία. Καταρχά, συμφωνώ με τον εισηγητή όσον αφορά ε, τον πολλαπλασιασμό των οικονομικών μέσων. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αρχίζει να βγαίνει πλέον από το δημοκρατικό μα έλεγχο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, οπότε συμφωνώ με αυτό το τμήμα τη έκθεση. Επίση, ε, αυτό που τονίζουν πολλοί συνάδελφοι ότι έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο εμπορικό ε, έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ε, νομίζω όμως ότι έχουμε τους πόρους να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε αυτό συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου Κάτι ακόμη το οποίο θα ήθελα να τονίσω και να προσθέσω ότι η προτεραιότητα για τον ενωσιακό προϋπολογισμό είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης εν μέρη χρειάζεται να το κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα μακροπρόθεσμο, μακροχρόνιο σχέδιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, με, ε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ετούντων άσυλο που φεύγουν από ζώνες ε, ε, εμπόλεμες. Πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες, τις εμπορικές στις διάφορες χώρες, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να ζητάμε λοιπόν μία αύξηση νομίζω για το, τις εμπορικές γραμμές ε, ως προς τα θέματα αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μονές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μούνιες. Συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέγκε, τον εισηγητή, όπω επίση και όλους όσου πήραν το λόγο για το θέμα αυτό. Δεν είναι μια πρώτη συζήτηση αυτή που κάνουμε σήμερα για το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστούμε για την γνωμοδότησή σας. Συμφωνούμε με κάποια από τα σημεία που έχετε αναφέρει. Κάποια από αυτά δεν εξαρτώνται τόσο από εμά, αλλά μπορείτε να μας έχετε εμπιστοσύνη, όσο, να, εμπιστοσύνη ότι θα τα διαβιβάσουμε στους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμών και κυρίως σε εκείνους που ασχολούνται με την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, και τα γενικά ζητήματα που θέσατε σε σχέση με τα καταπιστεύματα, τα trust funds. Όσον αφορά τώρα για τα, τα, τα θέματα που θέσατε για τα εμπορικά ζητήματα, πράγματι έχουμε έχουμε μια πολύ φιλόδοξη εμπορική ατζέντα και είναι γεγονός ότι μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν έχουμε αρκετούς πόρους για να τα υλοποιήσουμε. Όμως η αξιολόγησή μας, και αυτό φάνηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού ε, που υποβάλαμε στις αρχές του έτους είναι ότι οι πόροι που διατέθηκαν ε, στο σχέδιο προϋπολογισμού θα μπορούσαν να αντιστοιχούν ε, χονδρικά στις ανάγκες μας για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή αλλά και τις διαπραγματεύσεις των διαφόρων συμφωνιών που τις συνάπτουμε τώρα ή που ήδη τις εφαρμόζουμε, που ήδη ισχύουν. Καταλαβαίνουμε ότι το Trade for All, εμπόριο για όλους, είναι μια ανακοίνωση που αφορά ολόκληρες τις εμπορικές πολιτικές, όχι, όλες τις εμπορικές πολιτικές, όχι μόνο τη διαφάνεια και την επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν τις επενδυτικές πολιτικές. Όλα αυτά έχουν αποκρισταλωθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού ε, και μάλιστα είχαμε και μία συζήτηση με την Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών στις αρχές του έτους και είναι απολύτως ενήμερη για ε, τα όσα ε, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του Ιουνίου. Είναι περιορισμένος ο προπολογισμός μας, αυτό είναι αλήθεια, αλλά μπορούμε να έχουμε κάποια προγράμματα ε, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις διαπραγματεύσεις Κάποια από αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα η συμφωνία με την Νότια Κορέα και μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ε, καλύψουμε την επικοινωνία, τη διαφάνεια, ε, την κοινωνία των πολιτών ε, και όλες τις διαδικασίες, όλες τις δραστηριότητες επαφών και συνεργασίας δεν ε, μπορούμε να, ε, δεν είμαστε σε θέση να ζητήσουμε την εφαρμογή περισσότερων προγραμμάτων και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια το θέσαμε ως αίτημα στο, στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών ε, για τον προϋπολογισμό του έτους αυτού, του έτους αυτού. όμως τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εμπορική πολιτική δεν καλύπτονται από την επιχειρησιακό προϋπολογισμό μόνο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου αλλά και σε άλλες δημοσιονομικές γραμμές έχετε αναφέρει κάποιες από αυτές για παράδειγμα παράδειγμα το μέσο εταιρικής σχέσης, ε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων έχουμε κάποια μέτρα στην εμπορική πολιτική. Βλέπουμε, για παράδειγμα, την ανάπτυξη υποδομών στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών με τους εταίρους μας, αλλά και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό ισχύει κυρίως στο πλαίσιο του μέσου εταιρικής σχέσης, γιατί συνεργαζόμαστε ε, προκειμένου να υπάρχει ένα μέσο που θα διευκολύνει την εφαρμογή ε, της ε, του θεματολογίου μας για, την εμπορική, για, την, για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Αναφερθήκατε πολλές φορές στο θέμα της κυριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε να ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε όχι μόνο στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής αλλά και στο πλαίσιο πολλών προγραμμάτων που εφαρμόζει η DigiGrow όπως το COSME για παράδειγμα αλλά και σε προγράμματα όπως το μέσο εταιρικής σχέσης. Εν ολίγης θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός ε, αντανακλά τις ανάγκες αλλά και την ικανότητα που έχουμε στη γενική μας διεύθυνση να, ε, να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα και τα προγράμματα για να ε, μπορέσουμε επίσης να δώσουμε συνέχεια στην ανακοίνωση Trade for All με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Θα τις λάβω υπόψη. Θα ήθελα να ρωτήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η μελέτη για το μέσο της εταιρική σχέσης πότε θα είναι διαθέσιμη. Θα ήθελα να τη δω. ποιο θα είναι το περιεχόμενο, ποια θα είναι τα ποσά που θα αναφέρονται. Επίση, οι σημαντικές περικοπέ στη μακροοικονομική βοήθεια, που είναι σημαντικέ, αρκετά σημαντικέ. Μήπω θα μπορούσατε να μα δώσετε κάποιε εξηγήσει, αν όχι σήμερα, γραπτό κάποια στιγμή. Μπορούμε να λάβουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Ναι, για το θέμα του μέσου εταιρική σχέση, ναι, συγγνώμη, ξέχασα να απαντήσω τη σχετική ερώτηση. Αυτή η μελέτη δεν ε, είναι τίποτε το ιδιαίτερο. Είναι μία από τις αξιολογήσεις ε, που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εξωτερικά μέσα πολιτικών. Αυτό είναι ένα νέο μέσο, ε, το μέσο εταιρική σχέσης, οπότε πρέπει να περιμένουμε μία επιπλέον περίοδο εφαρμογής για να μπορούμε να κάνουμε μία εκ των προτέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων ε, που ε, ε, ε, υπήρξαν. Τα προβλήματα που είχαμε δει στο παρελθόν με παρόμοια μέσα δεν αφορούν κυρίως τα ποσά, αλλά τον τρόπο διεκπαιρέωσης των προγραμμάτων αυτών. Βλέπουμε την οικονομική διαχείρισή τους, για παράδειγμα, και ειδικότερα για το μέσο αυτό είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, γιατί η Γενική Διεύθυνση που, και, και η υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης που, έχει να, έχουν, που ασχολούνται με το ε, θέμα αυτό έχουν πολλά προβλήματα πόρων. Οπότε αυτό είναι το βασικό στοιχείο που θα εξεταστεί στην αξιολόγηση, αλλά θα δούμε και την εστίαση και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν ε, διεκπαιρεωθεί στο πλαίσιο του μέσου αυτού. Όσον αφορά την ερώτηση για τη μακροοικονομική ε, βοήθεια, ε, θα σας απαντήσω, βέβαια από κοινού, αφού συνεννοηθώ με τους συναδέλφους από την DJ ECFIN, για να είναι πιο ολοκληρωμένη η απάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ωραία. Η τροπολογία για την κατάθεση τροπολογιών για ε, το σχέδιο γνωμοδότησης 18 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Α, και θα ψηφίσουμε στις 31 Αυγούστου. Για να είμαστε έτοιμοι για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέργκε. Περνάμε τώρα στο σημείο 9. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κοινού κανόνες για τις εισαγωγές κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων από ορισμένε ε, τρίτες ε, χώρες, ε, γιατί από τη Λευκορωσία που δεν καλύπτονταν ε, γιατί κάποτε ήταν τμήμα της Ρωσίας ε, πρέπει να παίξουμε ε, ένα σημαντικό ρόλο με την επίλυση των συγκρούσεων στην Ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα στην περίπτωση της Ουκρανίας και θα συζητήσουμε για πρώτη φορά σήμερα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να ζητήσω πρώτον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει την παρουσίαση και επίσης έχω τη χαρά, νομίζω ότι για πρώτη φορά, να είναι εδώ ένα εκπρόσωπος τη δημοκρατία της Λευκορωσίας, ο κύριος Ρόμαν Σομπόλοφ, επικεφαλής ε, του Τμήματος Εξωτερικού Εμπορίου, τμήμα του Υπουργείου ε, Εξωτερικών ε, του, της Λευκορωσίας. Μετά θα σας δώσω το λόγο και για αυτήν την πρόταση, αλλά και ε, για τις εμπορικές μας σχέσεις. Να δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. My name is Mila. Καλημέρα σε όλους, λέγομαι Jeanne Mila από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, Trade, υπεύθυνη για τις εμπορικές σχέσεις με την Λευκορωσία. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, δεν μιλάμε συχνά εδώ στην Επιτροπή για τη Λευκορωσία, οπότε να σας κάνω μια επισκόπηση της κατάστασης για το εμπόριο και ευρύτερα για την πολιτική κατάσταση. Και μετά θα περάσω στην πρόταση της Κομισιόν λεπτομερέστερα. Κάποια στοιχεία. Σημαντικός εμπορικό εταίρο της Ένωσης η Λευκορωσία πέρυσι το 2015. Είχαμε δεκαδείς όγκο εμπορίου με την Λευκορωσία, 6 δις εξαγωγέ. Έχουμε λοιπόν πλεόνασμα εμπορικό 2 εκατομμύρια με την Λευκορωσία. Βελτιώνονται από το 14 σχέσεις μας, οι αμοιβέ. Είχαμε και θετικές εξελίξεις δηλαδή πιο ενεργό συμμετοχή της Λευκορωσίας στις εταιρικέ σχέσεις τις ανατολικές και είχαμε μια πιο επικοδομική τους στάση όσον αφορά την κρίση στην Ουκρανία. Ανάψη λοιπόν αυτών των θετικών εξελίξεων εξελίξαμε και εμείς ένα πιο έντονο διάλογο με τη Λευκορωσία και είχαμε στις 25 Φλεβάρου 16 ένα συμβούλιο υπουργών όπου αποφασίστηκε να αρθούν περισσότερε χειρός προς τη Λευκορωσία και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Λευκορωσία σε διάφορους τομείς. Αρρωγή, οικονομική, εμπόριο κλπ. Κύριος στόχος μας εδώ βέβαια είναι ο εξυγχρονισμός της οικονομίας της Λευκορωσίας προς όφελος και των Λευκορώσων αλλά και ημών μιας και είναι μεγάλος μας γείτονας. Τι κάνουμε συγκεκριμένα τώρα στο τομέα του εμπορίου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διαβούλευσης για τον εξυγχρονισμό της Λευκορωσίας είχαμε πιο έντονες ανταλλαγές σε σχέση με το εμπόριο και ξεκινήσαμε ένα εμπορικό διάλογο με την Λευκορωσία. Προχωράμε καλά. Θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση το φινόπορο και στόχος μας είναι να κάνουμε ανταλλαγές απόψεων για θέματα εμπορικά, ενδεχόμενες δυσκολίες και να δούμε Πώ το εμπορικό δίκαιο τέλο πάντων αναπτύσσεται, εξελίσσεται και στις δύο πλευρέ. Ένα σημαντικό στοιχείο στην εμπορική σχέση μα με Λευκορωσία είναι η, η προσχώρηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, κύριο στοιχείο για μα γιατί θα συμβάλλει στον εξυγχρονισμό τη οικονομία του. και θα μα επιτρέψει να του βοηθήσουμε μέσω διαφόρων προγραμμάτων για το capacity building όσον αφορά την προσχώρησή του στον ΠΟΕΠ. Από όλα αυτά ένα θα σας αναφέρουμε σήμερα. Αυτό που συζητήσαμε, που συμβάλλει δηλαδή στην ενίσχυση των εμπορικών μας σχέσεων με την Λευκορωσία. Δηλαδή η πρόταση για την κατάργηση ποσοστώσεων μονομερών όσον αφορά τα κλωστοφαρικά προέρχονται από τη Λευκορωσία. Να σας εξηγήσω κάπως τι είναι αυτός ο κανονισμός και τι θέλουμε να αλλάξουμε για να καταργήσουμε αυτές τις ποσοστώσεις που έχουμε τώρα με την Λευκορωσία. Αυτές οι μεμονωμένες ποσοστώσεις για την Λευκορωσία και τα κλωστοφερικά διέπονται από το 936-2015 και ένα κανονισμό της Κομισιόν, ένας εφαρμοστικός Κομισιόν και ένας χωριστός κανονισμός 2006 2015 οι ποσοστώσεις κλωστοεφαταρικών θεσπίστηκαν την 1η Γενάρη του 10 μετά την εκπνοή των διμερών συμφωνιών που είχαμε για τα κλωστοεφανταργικά που ανάγεται στο 93. Αν δείτε στις ποσοστώσεις έχουμε 21 κατηγορίες και αν δείτε την τωρινή χρήση αυτών των κατηγοριών θα παρατηρήσετε ότι είναι κάπως περιορισμένες, δηλαδή από τις 15 κατηγορίες για τις 15 από τις 21 η μέση χρήση μέσος όρος είναι γύρω στο 10%. Και μάλιστα υπάρχει μία κατηγορία η οποία χρησιμοποιείται ευρώς από την Λευκορωσία, η 117 κατηγορία, που αφορά φυσικές ίνες κλωστοφατουργίας, κυρίως μαλλί, οι οποίες τέλο πάντων έχουν πέρασει στην Ένωση. Αυτή λοιπόν η ποσόστοση χρησιμοποιείται κυρίως από την Λευκορωσία με ποσοστό 91% το 2014 και 99% το 2015. Περίπου δηλαδή 100% χρήση αυτής της ποσόστοσης. Θεωρούμε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις και ο αντίκτυπος της κατάργησης αυτών των ποσοστώσεων δεν θα έχει μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην Ένωση. Και ούτως ή άλλως παρακολουθούμε στενά το εμπόριο κλωσταφαντουργικών μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας. Βέβαια, αν κάτι πάει στραβά, έχουμε και άλλα εργαλεία να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν νομίζω τώρα να συμβεί και τίποτα. Εις βάρος δηλαδή της οικονομίας της Ένωσης. Συγκεκριμένα πάντως, τι προτείνουμε να αλλάξουμε στον τωρινό κατονισμό προτείνουμε να διαγράψουμε το παράρτημα 3, το παράρτημα δηλαδή ποσοστώσεων της Λευκορωσίας. Αυτή είναι η κύρια αλλαγή, γιατί δεν θα υπάρχουν πια ποσοστώσεις για τα κλωστοεφαντουργικά. Και επίσης, θέλουμε να κάνουμε κάποιες μικρότερες αλλαγές, εποφελούμε βέβαια τις ευκαιρίες, για να ρυθμίσουμε κάποια θέματα εναπομείναντα από τον κανονισμό. Έχουμε τη συνδυασμένη ονοματολογία στο παράρτημα 1 και επίσης θα βάλουμε και το επίσημο όνομα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στο παράρτημα 2. Γιατί αυτό που θα παραμείνει από αυτό το κανονισμό είναι οι ποσοστώσεις με τη Βόρεια Κορέα. Δεν έχουμε ποσοστώσεις για τα κλωστοεκτορικά με καμιά άλλη χώρα. Θα κάνουμε λοιπόν αυτή την προσαρμογή και θα αυξήσουμε την περίοδο ισχύω τη ε, έγκριση, τη άδεια από 6-9 μήνε. 6 μήνε είναι λίγο στενό σαν χρονικό διάστημα για την εφαρμογή. Και η τελευταία αλλαγή θέλουμε να αφαιρέσουμε πλήρως τις ποσοστώσεις για τη διακίνηση που αφορούν περισσότερο τις γειτονικέ χώρες. Ας πούμε όταν στέλνετε ένα μπλουζάκι στην Λευκορωσία τυπώνουν κάτι αυτοί και σας το ξαναστέλνουν. Ε, εντάξει, αυτό δεν ισχύει για την ε, Βόρεια Κορέα που είναι πολύ μακριά έτσι να στέλνουμε μπλουζάκια Οπότε και αυτό το τμήμα θα το διαγράψουμε. Αυτά από μένα. Και εδώ είμαστε. Δεν θα χαθούμε. Αν έχετε παραπάνω ερωτήσει. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Σόμπολεφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην Επιτροπή σας και για την ευκαιρία να μιλήσω στο τόσο εκλεκτό ακροατήριο. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια για τη σχέση μεταξύ Ευκορωσίας ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια είχαμε απτή πρόοδο όσον αφορά τις σχέσεις μας. Σήμερα οικοδομούμε μια οικονομική και πολιτική συνεργασία μέσω προγραμμάτων που θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ενός επικοδομητικού διαλόγου. Καλωσορίζουμε την απόφαση της Ένωσης του Φλεβάρου του Συμβουλίου για τη σχέση με τη Λευκορωσία και θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση ανοίγει νέες ευκαιρίες και νέα κεφάλαια για τη συνεργασία μεταξύ μας. Από το Φλεβάρι λοιπόν συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στις σχέσεις μας. Έχουμε και... Είχαμε και τον Απρίλιο του 2016 στις Βεξέλλες την ε, συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού Λευκορωσίας ΕΕ, την οποία χαιρετίζουμε και αυτό θα μας βοηθήσει περαιτέρω να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Είναι σημαντικό που αποφασίσαμε να διευρύνουμε το πεδίο διαλόγου μας στο, στον τομέα των τελωνίων, της ενέργειας, της γεωργίας. Στις 24 Μάη Επίσης είχαμε και, την, ε, και το φόρουμ στην Βιέννη όπου συμμετείχαμε και αυτό ήταν επιτυχές και θα μας βοηθήσει. Και βεβαίως όλα αυτά θα βοηθήσουν την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ Ένωσης και Λευκορωσίας. Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουμε βέβαια και διάλογο εμπορικό μεταξύ των ε, υπηρεσιών μας σε επίπεδο Υπουργείων και Γενικών Διευθύνσεων τη Κομισιόν, ώστε να δημιουργήσουμε μια μόνη πλατφόρμα διαλόγου για να διευκολύνουμε το διμερές εμπόριο και να άρουμε τους αναπομείναντες φραγμούς στις εμπορικές μας σχέσεις και να βελτιώσουμε βέβαια και το επιχειρηματικό κλίμα και να συμφίξουμε περισσότερο τις σχέσεις μας. Με την κατάργηση των μονομερών κυρώσεων θεωρούμε ότι έχουμε ένα πρώτο βήμα προς την άρση περί των φραγμών στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Λευκορωσίας και Ένωσης. Όπως ξέρετε, από το 1993, εδώ και πολύ καιρό δηλαδή, είχαμε συμφωνία εμπορική μεταξύ Λευκορωσίας και Ένωσης μέχρι το 2010, όπου είχαμε τη διμερή συμφωνία για το εμπόριο και τα κλωστεφερικά προϊόντα. Έχουμε αυτά λοιπόν τα προϊόντα που φτάνουν στην Ένωση. Είχαμε περιορισμούς που είχαν καθοριστεί για 34 κατηγορίες από τις 164 κατηγορίες λευκορωσικών κλωστοεφαντουργικών. Το 2008 είχαμε επαφές μεταξύ Λευκορωσίας και Κομισιόν και ως συνέπεια καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις για 13 από 33 κατηγορίες, κατηγορίες το 2009 και από το 10, το Ιανουάριο του 10 ευθέτησε απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση για μονομερείς ποσοστό όσον αφορά τι ε, εξαγωγέ κοστοφορικών από Λευκορωσία στην Ένωση. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η απόφαση για την θέσπιση των, των ε, ποσοστών από το 10 μονομερό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν βασίζεται σε διμερεί ε, συμφωνίε, διεθνεί συμφωνίε με τη Λευκορωσία. Οι μονομερεί λοιπόν ποσοστώσει για αυτέ τι κατηγορίε λευκορωσικών προϊόντων αντικατέστησαν τη συμφωνία που δεν μπορέσαμε να ανανεώσουμε μετά το 2010 και μετά την προσχώρηση στην Ελληνική Ένωση της χώρας μας με την Ρωσία και το Καζακστάν. Τα κλωστοβατρικά μας λοιπόν θα φτάσουν στην αγορά της Ένωσης και αυτά, αυτό θα αφορά τα προϊόντα μας ανεξάρτητα από την προλεύσή του και τον τρόπο μεταφορά τους. Πάντως αυτά που έχουν γίνει αποδεικνύουν ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η Λευκορωσία απέχει πολύ από την χρήση, την πλήρη χρήση ποσοστώσεων σε 21 κατηγορίες και όπως είπε η Κομισιόν, το 2015 χρησιμοποίησαμε κατά μέσο όρο της ποσοστός από 1 μέχρι 16% εκτός από τα κλωστοφαρικά λίνου. Για την πλειοψηφία των κατηγοριών ο μέσος όρος χρήσης είναι γύρω στο 10%. Η περιορισμένη λοιπόν χρήση αυτών των αυτόνομων ποσοστώσεων στην εισαγωγή των κλωστοφατορικών σημαίνει ότι έχουμε πολύ περισμένο αντίκτυπο στο εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες εργάζονται στον τομέα της κλωστοφατορικής Λευκορωσία είναι ιδιώτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει επαγγελμένες επαφές μεταξύ των προσώπων των δύο πλευρών. Πάντως αυτές οι σωστώσεις δεν ευνοούν τη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και θα πρέπει να πούμε ότι η Λευκορωσία ως άμεσος γείτονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μόνη χώρα, η δεύτερη μαζί με την μάλλον ε, Βόρειο Κορέα, όπου υπάρχουν ποσοστώσεις για αυτά τα προϊόντα. Και αυτό είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανεί από τη στιγμή που δεν βρισκόμαστε στον κατάλογο μεγάλων παραγωγών κλωστοφαντουργικών. Βεβαίως ο λόγος πίσω, μάλλον που διέπει αυτές τις ποσοστώσεις είναι οικονομικός. Θεωρούμε ότι οι θετικές εξελίξεις της σχέσης μεταξύ Ένωσης και Λευκορωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και επίσης η Λευκορωσία να σας πω σε αυτό το θετικό υπόγραφο, προτείνει την κατάργηση αυτών των ποσοστώσεων για όλα τα κλωσταφατικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη Λευκορωσία. Πρέπει επίσης να πούμε ότι στις 9 του Ιούνιου του 2016 στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραγωγών Κλωστοβαρχικών Προϊόντων έγινε δεκτή η Ομοσπονδία, η Λευκορωσική Ομοσπονδία Κλωστοφαρουργών ως μέλος. Και υπόθηκε ότι θα πρέπει να αρθούν αυτές οι κυρώσεις και περιορισμοί κατά των λευκορωσικών προϊόντων. Συνοψίζοντα, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, συνεργασία μα ώστε να βελτιωθεί, βρεθούν οικονομικέ συνθήκε αμοιβέ και η συνεργασία μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για μα όσον αφορά στι εξαγωγέ μα. Στόχο τη τωρινή μα πολιτική είναι να διαφοροποιήσουμε τι εξαγωγέ μα και γι' αυτό ακριβώ το λόγο ε, θεωρούμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι των εξαγωγών μα θα πηγαίνει στην αγορά τη Ένωση. Και η άρση των κυρώσεων βεβαίω θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προ αυτή την κατεύθυνση και θα στείλει ένα σημαντικό μήνυμα στι επιχειρηματικέ κοινότητε και στις δύο πλευρέ. Είμαι πεπισμένο ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις σε μια αμοιβαία κοινοφελή βάση και στην εξυπηρέτηση των αμοιβαίων συμφερόντων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε ερωτήσει, ευχαριστώ να τι απαντήσω. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Σομπόλιεφ για την ε, συμβολή σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε από το Μίνσκ εδώ στην Επιτροπή μας που κάνατε τόσο δρόμο. Και αν έχετε ερωτήσεις, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά θα δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Σομπόλιεφ. Πρώτα ο συγκητής μας, ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως συζητητής για το θέμα αυτό, Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση της Επιτροπής καθώς και την παρέμβαση του κυρίου Τσόμπολιεφ. Αυτή η πρόταση, ίσως περισσότερο από άλλες που συζητάμε, αποδεικνύει ότι το εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι βασικό τμήμα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μας. Την προώθηση δηλαδή βασικών μας αξιών στον κόσμο. Οι σχέσεις ε, Ένωσης Μπελαρούς έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, συνεχίζουν να βελτιώνονται. Αυτό είναι καλό για αμφωτέρους. Η Μπελαρούς είναι ε, εν δυνάμει στρατηγικός μας εταίρος έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει για την προσπάθεια διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση συγκρούσεων στην ανατολική μας γειτονία. Θα μπορούσε να είναι γέφυρα μεταξύ της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ευρωρωσικής Οικονομικής Ένωσης, της οποίας είναι μέλος. Πιστεύω ότι μια ενιαία περιοχή εμπορίου από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαντιβοστόκ μπορεί να βοηθήσει. Είναι μεν δύσκολη σε αυτή τη συγκυρία, αλλά πρέπει να είναι πάντα μακροπρόθεσμος στόχος. Η οικονομική επίπτωση της πρότασης της Κομισιόν είναι αμελη, ε, γιατί δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες. Πρέπει να θεωρηθεί ως τμήμα ενός πακέτου που θα βοηθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη των σχέσεων Ένωσης Μπελαρούς. Και θα ήθελα να ενθαρρύνω την Μπελαρούς να προωθήσει τις σχέσεις ένταξης των ΠΟΕΡ που γίνονται χωρίς μεγάλη πρόοδο εδώ και 23 χρόνια. Είμαι πεπισμένος ότι η συμμετοχή στον ΠΟΕ θα παρήχε πολλές περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του εμπορίου της Μπελαρούς και άρα ανάπτυξη και της ευημερίας της χώρας. Ευχαριστώ πολύ και ε, να ακούσω τώρα και τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων μας. Να δώσω το λόγο στους Κιώδης. Πρώτος ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητά συγγνώμη η Ιτσίκου δεν είναι παρόν γιατί είχε ορισμένες υποχρεώσει στην εκλογική του περιφέρεια και δεν μπορεί να παρευρεθεί. Μου ζήτησε λοιπόν να σας διαβάσω το εξής κείμενο. Είμαι θετικό έναντι τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τροποποιηθεί ο κανονισμό 2015-1936 για τι αγωγέ εκλώσεων ευρωδικικών από ορισμένε τρίτε χώρε. Η απελευθέρωση στι 22 Αυγούστου 2015 όλων των πολιτικών κρατουμένων στην ε, Μπελαρού ήταν ένα βήμα που το είχε ζητήσει επανειλημμένα και το ανέμενε από καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονό ε, αυτό είχε μεγάλη σημασία και το αντιμετωπίσαμε αισιόδοξα ως Κοινοβούλιο. Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Μπελαρού στα τελευταία δύο χρόνια. Συμμετέχει ενεργά στην ε, ανατολική εταιρική σχέση, προωθεί τον εξυγχρονισμό της, συμμετέχει σε προγράμματα όπως το Erasmus και σε προγράμματα ανταλλαγών για τις βέλτιστες επιστημονικές πρακτικές. Όλα αυτά είναι μηνύματα που φαίνεται ότι ε, αρχίζει μία προσέγγιση της Μπελαρούς προς τις αξίες της ε, Ευρώπης, αν και γίνεται με αργό τρόπο και με δυσχέρειες αυτή η προσπάθεια. Άρα οι αυτόνομες προσωστώσεις για τα κλωστοφαντουρικά και τα ενδύματα είναι σημαντικό μήνυμα για να αναπτυχθούν οι σχέσεις που δεν πρέπει να βασίζονται μόνο σε απλώς εμπορικά συμφέροντα. Βεβαίως, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και η κατάργηση της θανάτικης ποινή είναι πλευρές που μας ανησυχούν ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θέλουμε σύντομα δείγματα ότι θα, θα αλλάξει η κατάσταση για αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα εν ώψη των εκλογών του προσεχούς φθινοπόρου, που θα είναι σημαντικό σημείο, σταθμός για να σημειωθεί πρόοδος. Η ομάδα μου θα να στηρίξει αυτή την πρόταση. Και επειδή η κατάργηση των δασμών για τα προϊόντα αυτά θα έχει περιορισμένη επίπτωση στην εσωτερική αγορά, αλλά γιατί έχει έννοια σε ένα πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου ο σεβασμός της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η περισσότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Οι σοσιαλιστές, η Καρολίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτά που ακούσαμε οι εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεργασία με την Μπελαρούς είναι σημαντικό μήνυμα και είναι σημαντικό να δούμε συγκεκριμένα, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχουν βελτιώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι αποφασιστικό για την κατάργηση αυτών των ποσοστώσεων. Βλέπουμε αξιοσημείωτες και απτές θετικές εξελίξεις. Έχουμε τις εκλογές τον, το Σεπτέμβριο Εκεί θα φανεί αν οι εξελίξεις θα πάνε προς θετική κατεύθυνση και αυτό θα είναι το αποφασιστικό και τη δική μου απόφαση. Για το θέμα αυτό να προσθέσω ακόμη ότι συμφωνώ από τεχνική πλευρά όντως αυτές οι ποσοστώσεις ή μάλλον η κατάργησή τους ε, δεν θα δημιουργήσουν μεγάλες αλλαγές. Γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαν καν εξαντληθεί αυτές οι ποσοστώσεις. Αλλά είναι σημαντικό μήνυμα ότι κάνουμε κάτι για να το δει και η Μπελαρούς ότι τους δίνουμε δυνατότητες βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων και είναι επίσης ένα σαφές μήνυμα ότι αναγνωρίζουμε τις θετικές εξελίξεις. Όπως υπόθηκε ε, με ενδιαφέρουν οι εκλογές και θα ήθελα να δω τι θα πούν και οι παρατηρητές μας που θα συμμετάσχουν στις εκλογές και βεβαίως έχουμε και μια ειδική ομάδα εργασίας για τη σχέση με την όπου μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά τα θέματα αυτά και μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Υπάρχουν μέτρα προστασίας. Υπάρχει αυτή, αυτό το καθεστώς παρατηρητή. Τι θα γίνει αν ε, στο μέλλον επιδενωθούν οι σχέσεις ε, εφόσον θα έχουμε καταργήσει τις ποσοστώσεις. Θα ήθελα να μπορέσουμε να δούμε συγκεκριμένα τι γίνεται. ούτως ώστε αν ε, σημειωθούν θετικές εξελίξεις και τις διαπιστώσουμε, ε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Χαίρομαι για τη συνεργασία και ευχαριστώ τον κύριο Τάκουλα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάμπ. Ευχαριστώ. Εμείς το ECR καλωσορίζουμε αυτά τα βήματα από τη Λευκορωσία για την ε, απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και την ε, βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι είναι καλό το ότι πηγαίνει πιο, προς πιο ε, διεθνώς αποδεκτές δημοκρατικές προδιαγραφές και πρότυπα. Εγώ μέχρι στιγμής προσπάθησα να μην συνδυάσω πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα με το εμπόριο. Νομίζω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι που αντιμετωπίζεται σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο, γιατί το εμπόριο ε, πολλές φορές ε, προσπαθώντας να αυξήσει την ευημερία δημιουργεί προβλήματα στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις. Πρέπει να πω βεβαίως ότι στην ομάδα μας υπάρχουν αντιπροσωπείες που έχουν σοβαρές ανησυχίες ε, για τη Λευκορωσία και πιστεύουν ότι οποιασδήποτε παραχωρήσεις πρέπει να συνδεθούν με την, τον περιορισμό των, της νοθείας στις εκλογές. Ε, αυτό λέω αυτό εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν στις 11 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας ε, για αυτήν τη σύνδεση με τις ε, εκλογικές απάτες. Ελπίζουμε να μην οδηγήσουν τη Λευκορωσία προς την κατεύθυνση της Μόσχας και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις εκλογές και να, υπάρξουν, να υπάρξει εκλογική αναμέτρηση που θα χαρακτηρίζεται λιγότερο από την απάτη. Ευχαριστώ πολύ. Για ε, την δεν έχουμε σκιώδη γιατί αλλά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σόλτς. εγώ ευχαριστώ τον συγητή για αυτήν την εισαγωγή. Αλλά να αναφέρω ένα πρόβλημα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες θέλουμε να υπάρχουν ε, πολύ σαφείς ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βιώσιμης ανάπτυξης. Τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να παρακολουθούμε μετά και την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών. Αυτό πρέπει να αναφερθεί όταν συζητάμε και για την κατάργηση ποσοστώσεων και γενικά για τη διαμόρφωση των εμπορικών σχέσεων με την Πελαρούς. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν ε, είναι σωστή η διατύπωση που λέμε ότι θέλουμε να εφαρμοστούν παγκόσμια οι ευρωπαϊκές αξίες. Εμείς θέλουμε με τις εμπορικές μας σχέσεις να συμβάλλουμε ούτω ώστε σε κάθε χώρα οι δημοκρατικά εκλεγμένοι να εφαρμόζουν δημοκρατικές αξίες, να συζητούν ανοιχτά με την κοινωνία να, και μετά να γίνεται σεβαστή νομοθεσία. Αυτό μπορούμε να πούμε σε μια διμερή εταιρική σχέση. Να συμβάλλουμε δηλαδή, ούτω ώστε να υπάρχουν προδιαγραφές για κοινωνικά θέματα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό η ομάδα μας διαπιστώνει συγκεκριμένες προόδους στην εσωτερική εξέλιξη της Μπελαρούς, αλλά ε, αυτή η διατύπωση ότι η αλλαγή θα έρθει μέσω του εμπορίου είναι συζητήσιμη. Βεβαίως, μπορούμε να ασκήσουμε πίεση, αλλά δεν θα πρέπει να είναι η μόνη μας ε, δυνατότητα δράσης. Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις σχέσεις μας με διάφορες χώρες. Άκουσα όλα αυτά που υπόθηκαν Θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να δούμε πώς ακριβώς πρέπει να τροποποιήσουμε την έκθεση, τι πρέπει να προχωρήσουμε και φυσικά οι εκλογές είναι σημαντικό γεγονός και θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε. Πριν δηλαδή διαμορφώσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας και στον εμπορικό τομέα. Κάτι άλλο που δεν πρέπει να, ξεχνά, να ξεχνάμε γιατί είχαμε την επέτειο του Τσερνόμπιλ φέτος. Ε. Είναι 40 χρόνια. Η προσοχή στα οικολογικά θέματα πρέπει να είναι σημαντικό στοιχείο των σχέσεών μας. Θα έπρεπε να μας ενημερώσει η Μπελαρούς σε τι βαθμό έχει ε, εφαρμόσει τις διεθνείς συμφωνίες για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μπούχνερ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίασή του και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Σόλτς μόλις τώρα. Η ομάδα μου και εγώ προτείνουμε να περιμένουμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές στις 11 Σεπτεμβρίου και να έχουμε πρώτη αποτίμηση για το πώ διεξήχθησαν. Δεν είναι και ουσιώδης καθυστέρηση. Ούτω η έκθεση θα ψηφιστεί το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, συγγνώμη. Από τότε που ήρε το Συμβούλιο τη Κυρώσης, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει σημειώσει μεν πρόοδο, αλλά σίγουρα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που θα θέλαμε. Οι αρχές της ε, Μπελαρούς είχαν τις συγκεκριμένες ε, προτάσεις του ΟΣΑ για την προεδρική εκλογή, αλλά τις εφάρμοσαν μόνο εν μέρη. Επίσης οι αρχές της χώρας δεν έχουν εγγυηθεί τα δικαιώματα πολιτικά και κοινωνικά των πρώην πολιτικών κρατουμένων και δεν έχουν γίνει επίσημα θεσμικά βήματα για να εγγυηθούν ε, την ελευθερία του συνέρχεσθε και η συνεργασία τους με τον εισηγητή τον, του ΟΗΕ δεν είναι πλήρης. Αναφερθήκαμε ήδη στη θανατική ποινή, δεν έχει ακόμη καταργηθεί. Φέτος εκτελέστηκαν ήδη τρεις θανατικές πηγές, ε, ποινές, συγγνώμη. Συγγνώμη, επιβλήθηκαν, δεν ξέρουμε αν έχουν ε, εκτελεστεί. Οι εκλογές 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα είναι ε, ένα σημαντικό γεγονός για την Λευκορωσία. Να δούμε ε, αν θα σταματήσει η μακρόχρονη παράδοση νοθείας στις εκλογές. Και ελπίζουμε οι αρχές να αντιμετωπίσουν θετικά τους πολίτες της χώρας και τις σχέσεις τους με την Ένωση. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, αλλά θα ήθελα την επιβεβαίωση πριν βελτιώσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με την Λευκορωσία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάτμοφ. Ντάτμουθ, εμένα είπατε. Α, ευχαριστώ πολύ. Το άκουσα αλλιώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρειάζεται να επαναλάβουμε, πιστεύω, ότι όπως διαβάσατε σε εφημερίδες έγινε ένα δημοψήφισμα στι ΗΠΑ που κατέληξε με κάποιο τρόπο. Αλλά θα πρέπει να ξαναπούμε που, κάτι που είπε τόσο εύγλωτα ο Ντόναλτ Τούσκ ότι μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύεται από όλου του συνοσιακούς κανόνε και θα συνεχίσει να συμβάλλει και στον προπολογισμό. Οπότε έχει έννοια η συμμετοχή μα. Θα προτιμούσα να μην έχει ημερομηνία λήξη, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Σε σχέση με αυτά που είπε ο εισηγητή. και αυτά που είπαν οι συνάδελφοι Γκουε και Πρασίνων. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι κάτι που πάντα είναι έμεσο στοιχείο της εμπορικής πολιτικής είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θεωρεί μηχανισμό για να προωθήσουν, όπως λέτε, ευρωπαϊκές αξίες και για να, χρησιμοποιήσουν, να τις χρησιμοποιήσουν ως ε, ένα όργανο της εξωτερικής πολιτικής. Άρα το εμπόριο δεν είναι στην ουσία θέμα εμπορίου, δεν είναι κυρίως καν θέμα εμπορίου η εμπορική πολιτική δηλαδή της Ένωσης. Και αυτά που είπε ο εισηγητής και ο κύριος Σόλτς και ο κύριος Μπούχνα, τον οποίο καλωσορίζω, αν και δυστυχώ δεν είναι πια εδώ να ακούσει το καλωσόρισμα, όλοι κατέστησαν απόλυτα σαφές, απόλυτα σαφές, 1000% σαφέ ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να χρησιμοποιηθεί και θεωρείται μηχανισμός προώθηση στόχων εξωτερική πολιτική. Αυτό δεν είναι προ το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε της Ένωση, ούτε του εμπορίου. Και είναι κάτι για το οποίο λυπάμαι ιδιαίτερα και με το οποίο είμαι εντελώ αντίθετο. Και δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο εγώ επινοώ, είναι κάτι που υπόθηκε εκπεφρασμένα. Και κάτι άλλο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν για την κατάργηση αυτών των ποσοστώσεων για τα κλώστο ή Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει αναλύσει τα στοιχεία η για το γεγονός ότι σε χώρες της Ένωσης όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία έχουμε ισχυρό κλωστιφαντουργικό κλάδο. Και τι βλέπουμε να έχει συμβεί. Ο δικός μας κλάδος στην Ένωση δεν συμφωνεί με την κατάργηση των ποσοστώσεων. Και πραγματικά πέστε μου πώς αναλύετε την κατάσταση. Ε, την έχετε αναλύσει καθόλου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να περάσουν από το Συμβούλιο, ούτε καν από το Κοινοβούλιο. Ίσως θυμούνται ορισμένοι συνάδελφοι την επίγουσα βοήθεια για το Πακιστάν μετά από πλημμύρε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Η πρόταση που ήταν βεβαίως λογική πρόταση από τη Βρετανική κυβέρνηση που συνήθως αυτά που προτείνει δεν περνάνε από το Συμβούλιο. Είπαν ότι θα έπρεπε να μειωθούν οι δασμοί και να αυξηθούν οι ποσοστώσεις εξαγωγών του Πακιστάν, ιδιαίτερα να μειωθούν να γίνουν αυτά γενικότερα για τα κλωστεφαντουργικά και διαπιστώσαμε ότι για να περάσει αυτή η πρόταση πέρασαν τρία χρόνια. Ε, σε τρία χρόνια μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι οι επιπτώσεις ε, από τις πλημμύρες είχαν αντιμετωπιστεί. Οπότε η ερώτησή μου, κάνατε ανάλυση και απευθύνεται προς την Κομισιόν, κάνατε ανάλυση για το πώς όσοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των δικών μας κλωστοεφαντουργικών προϊόντων και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο θα αντιδράσουν. Τι ανάλυση κάνατε και τι αποτελέσματα είχε. Και επανέρχομαι σε κάτι που επανειλημμένα έχω πει. Και στο βιβλίο που όποιο θέλει μπορώ να του δώσω αργότερα, αναφέρω ότι είναι πιο δύσκολο να υπάρξει εμπορική συμφωνία όταν έχει 28 χώρε από ότι είναι αν ήταν μόνο μία χώρα. Και αυτό καταδεικνύει η πείρα της Ελβετίας και άλλων. Δεν είναι ευκολότερο, είναι δυσκολότερο. Το BBC θα σας πει αυτές τις βλακίες ότι είναι τόσο εύκολο ε, γιατί είναι ένα μεγάλο μπλοκ. Καθόλου δεν είναι πιο εύκολο. Και ναι μεν ε, ε, υπήρξα ιδιαίτερα επικριτικός έναντι της Επιτρόπου Εμπορίου Σεσίλια Μάλστρομ. Αναγνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο καθήκον να συνδυάσεις τα συμφέροντα 28 χωρών, 28 οικονομιών που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από πλευράς ε, διάρθρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Στρέφουμε τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως ο κύριος Σομπόλεφ μπορεί να πάρει το λόγο μετά, αν το επιθυμεί. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω πρώτα τις τεχνικές ερωτήσεις και μετά τις πιο πολιτικές. Το πρώτο ερώτημα ήταν τι θα συμβεί αν δούμε σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις αγορές της Ένωσης λόγω της κατάργησης αυτών των ποσοστώσεων, προφανώς έχουμε ακόμη τη δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να επαναφέρουμε τις ε, ποσοστώσεις, ε, πάντοτε έχουμε τη δυνατότητα νομικώς να το κάνουμε αυτό, ε, όμως δεν λέω ότι αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ένα καλό και εύρυθμο μηχανισμό παρακολούθηση του πώς λειτουργεί το σύστημα, έχουμε ρήτρε ε, ε, διασφάλισης ε, για να δούμε τι θα συμβεί αν υπάρξει κάποια ζημιά. Υπάρχουν λοιπόν πολλούς τρόπους να αντιδράσουμε αν συμβεί κάτι το αρνητικό και θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι ότι θα μπορεί η Λευκορωσία να εξάγει τα κλωστοεμφαντουργικά της προϊόντα χωρίς ε, κανέναν έλεγχο. Μιλάμε για 8 με 20%. Δεν είναι ότι είναι απολύτως ανοιχτή η αγορά, εντελώς ανοιχτή. Ε, ε, θα έχουμε και κάποιους δασμούς ακόμη, κάτι το οποίο μας αποφέρει έσοδα. Το ερώτημα τώρα είναι κατά πόσο αν έχουμε κάνει λεπτομερή ανάλυση για τον αντίκτυπο της κατάργησης των ποσοστώσεων αυτών ε, στην αγορά της Ένωσης ε, και στον κλάδο των, ε, της κλωστοϊφαντουργίας της Ένωσης. Κοιτάξτε, δεν έχουμε μία μελέτη όντως εκπονήσει, γιατί πιστεύουμε επειδή είναι μικρός ο όγκος ο εμπορικός, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο και Ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό, οπότε προσπαθούμε να εστιαστούμε ε, ε, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι ε, είχαμε πολύ μακροχρόνιες συζητήσεις και στο Συμβούλιο, στην αρμόδια, ομόδια, στην αρμόδια ομάδα εργασίας που αφορούσε ακριβώς την κλωστοϊφαντουργία. Ήταν δηλαδή εκεί επιρρογνώμονες του κλάδου, μιλούμε με τον κλάδο κάθε μέρα, έχουμε επαφές μαζί του ε, και έχουμε πολλές ομάδες που το εξετάζουν. Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ε, δεν θα αρχίσουμε τώρα να ανοίγουμε ιστορίες χωρίς ε, λόγο. Έχουμε ένα σύστημα, ένα μηχανισμό διασφαλίσεων, αν παρά το ότι έχουμε κάνει όλη αυτή την εργασία υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος για το ερώτημα που αφορά τώρα το κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ της πρότασης αυτής ε, και των ε, προσεχών εκλογών στη Λευκορωσία. Επισήμως από πλευράς μας όχι. Αλλά όπως ανέφερα και στην ε, εισαγωγή μου, ε, είναι τμήμα μιας ευρύτερης πολιτικής διαδικασίας ε, συνεργασίας ε, με την Λευκορωσία. Τώρα οι συνάδελφοι, οι αρμόδιοι συνάδελφοι από την Επιτροπή, εσείς και το Συμβούλιο, επίσης έχετε κάποια συμμετοχή σε αυτό. Είναι τμήμα μια ευρύτερης διαδικασίας, πράγματι. Εγώ προσωπικά, που δεν είμαι βέβαια εμπειρογνώμονας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν ας πούμε τη Λευκορωσία και πολλές άλλες ε, χώρες ε, γειτονικές μας ε, δεν νομίζω ότι είναι μια χώρα που θα έπρεπε να με την οποία θα πρέπει να σταματήσουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές. Υπάρχουν άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Για μένα λοιπόν δεν είναι θέμα αυτό. Και για να αναφερθώ στο τελευταίο ερώτημα του κυρίου Τάρτμουθ, ε, για το κατά πόσο είναι ευκολότερο να συναυθεί μια εμπορική συμφωνία με 28 χώρες ή με μία. Εγώ συμμετείχα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση της Τρογγυλής Τράπεζας ε, στις 21 Ιουνίου στο Κοινοβούλιο, η οποία αφορούσε μια μελέτη και μια ανάλυση που είχε γίνει νομίζω από ένα οικονομικό Ινστιτούτο στην Αυστρία για ακριβώς αυτό το θέμα, τι είδους διμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες ε, υπάρχουν και αφορούσε ε, την ΕΦΤΑ ε, θα σας ε, συμβουλεύσω να διαβάσετε αυτήν την μελέτη γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κύριε Σομπόλεφ, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, γνωρίζετε η Λευκορωσία ήταν βασικό θύμα, κύριο θύμα της καταστροφής του Τσερνομπίλ. 30% της επικράτειάς μας υπέστη το τεράστιο αυτό το πρόβλημα. Για μας λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι πληρούμε όλες μας τις ε, ε, υποχρεώσεις, ότι τις εκπληρώνουμε όλες μας υποχρεώσεις προς τον τομέα αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση για το θέμα αυτό. Ε, σεβόμαστε όλες, μας, όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε ως προς τα περιβαλλοντικά. Όσον αφορά τώρα τη σχέση μεταξύ των εμπορικών ζητημάτων, ειδικότερα ε, της κλωστοεφαντουργίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και όσον αφορά την θανατική ποινή Προφανώς ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει αν θα κάνει αυτή τη σύνδεση, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ε, δύο μέτρα και σταθμά. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε την τελική εκδοχή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ε, στην οποία επίσης υπάρχει ακόμη η θανατική ποινή. Για μένα θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω κατά πόσο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν την υποχρέωση να καταργήσουν θανατική ποινή στο πλαίσιο της ε, συμφωνίας αυτής. Ε, αυτές, αυτοί οι περιορισμοί, τέλος πάντων όχι περιορισμοί, αλλά οι ποσοστώσεις αυτές, δεν επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον όγκο του εμπορίου της χρωστοεφαντουργίας μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λευκοκολοσία, ειδικότερα για τα ενδύματα, η κατάργηση αυτή θα είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα, όχι μόνο προ ε, την κυβέρνηση τη Λευκορωσία και τι κυβερνήσει των κρατών μελών, αλλά θα είναι και ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα προ την επιχειρηματική κοινότητα ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, μπορείτε να κάνετε εμπόριο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα νέο επίπεδο προετοιμασίας που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στάκουλα, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα λοιπόν και εγώ να κάνω τα καταληκτικά μου σχόλια στην υπέροχη γλώσσα μου τα φινλανδικά. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν τις απόψεις τους και συνέβαλαν στη συζήτηση. Νομίζω με καλή συνεργασία θα είναι πολύ καλό και το αποτέλεσμα, μια πολύ καλή έκθεση και νομίζω ότι είναι κοινό το συμφέρον μας η ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας. Θέλουμε να την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει προς το, προς την πορεία της προς τη δημοκρατία. Τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το θέμα της θανατικής ποινής ε, βεβαίως ε, Συμφωνώ με αυτό που μόλις είπε ο κύριος Σοβόλεφ ε, εκ μέρους της Λευκορωσίας και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους με τον ίδιο τρόπο και πρέπει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θανατικής ποινής πρέπει βεβαίως να το αντιμετωπίσουμε. Ε, έχει να κάνει με τη σχέση μας ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Ιαπωνία και κάποιες αραβικές χώρες που ακόμη επιβάλλουν τη θανατική ποινή. Πρέπει λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε όλες τις χώρες αυτές που ακόμη επιβάλλουν τη θανατική ποινή με τον ίδιο τρόπο. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις μας, εγώ πιστεύω ότι η Λευκορωσία μπορεί να μας, να δείξει το δρόμο στις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα, πώς μπορούν και εκείνες να ξεφορτωθούν τη θανατική ποινή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως να μην έχουμε δύο, και, δύο μέτρα και δύο σταθμά, και να αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όλες τις χώρες. Επίσης, χρειαζόμαστε και έναν πρωταθλητή ε, αξιών ε, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας έκφρασης, που είναι οι βασικές ε, θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα εκπονήσω την έκθεσή μου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ελπίζω ότι όταν θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβρη θα μπορέσουμε να το εξετάσουμε μετά τις ε, εκλογές στη Λευκορωσία και ελπίζω ότι μετά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ε, σε πολύ θετικό πνεύμα και να προχωρήσουμε ε, τη συνεργασία μας με αυτόν τον πολύ σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε θα μπορέσει να καρποφορήσει. Αυτά για την ώρα από πλευράς μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα την, ε, ε, τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής μας ε, για να μπορέσω να διαμορφώσω ε, τη συμφωνία αυτή ώστε να μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές ε, ως προς την προβολή των ευρωπαϊκών αξιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στις 31 Αυγούστου και θα ψηφίσουμε στις 26 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικότερα τον κύριο Σομπόλευ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επτά λεπτών και μετά θα αρχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών.